Uh, good morning, ladies and gentlemen. Please take your seats. Uh, I don't know where more. Λοιπόν, δεν ξέρω που είναι περισσότεροι συνάδελφοι, λέει ο πρόεδρος Αλλά ας υποθέσουμε... Ας υποθέσουμε ότι κάπου εδώ θα είναι. Όπως θα έλεγαν οι επιστήμονες στα πειράματά τους. Σήμερα έχουμε το σημείο 10 στην ημερήσια διάταξη το οποίο αποφασίστηκε χτες για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την κινητικότητα και τις μεταναστεύσεις και τη σχέση τους με τα εσωτερικά χρηματοδοτικά μέσα. Έχουμε επίσης και μία παρουσίαση από την Διεθνή Οργάνωση Μετανάστευσης, την οποία εκτιμάμε ιδιαίτερος για αυτά τα οποία έχουν κάνει και από την οργάνωση Concord, μια οργάνωση πάρα πολύ σημαντική. Θα ξεκινήσουμε με την ανταλλαγή απόψεων. Λοιπόν, όπως γνωρίζετε, το Νοέμβριο Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανακοίνωση για τη συνολική αντιμετώπιση της μετανάστευσης και της κινητικότητας. Έχει τέσσερις πυλώνες η ανακοίνωση της Επιτροπής. Νόμιμη μετανάστευση και κινητικότητα, παράνομη μετανάστευση και σωματεμπορία, διεθνής προστασία, πολιτική ασύλου και τέλος μεγιστοποίηση των αναπτυξιακών συνεπειών της μετανάστευσης και της κινητικότητας. Υπάρχει και ένα κείμενο εργασίας που ονομάζεται «Μετανάστευση και Ανάπτυξη», το οποίο θέτει, θα έλεγα, τα θέματα τα οποία συνδέουν τη μετανάστευση και την αναπτυξιακή πολιτική. Αυτό το θέμα παρουσιάζει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους ε, φορολογουμένους μας, οι οποίοι μας ζητούν γιατί ξοδεύω τόσα πολλά χρήματα ε, σε άλλες χώρες. Ε, τι έχω να κερδίσω από αυτό, τι κερδίζουν αυτές οι χώρες. Πέρα από το ηθικό το θέμα βέβαια, θέλουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, ο οποίος ζει σε ένδια και σε στερήσεις και στη δική μας χώρα όμως και στις δικές μας χώρες συμβαίνει αυτό. Προσπαθούμε να σταματήσουμε τη μαζική μετανάστευση, αντιμετωπίζουμε το θέμα της μετανάστευσης λόγω των κλιματολογικών συνεπειών. Πρόσφατα είχα πάει στην και μου είπε ο Πρωθυπουργό της χώρας ότι ανεβαίνουν πάλι τα επίπεδα των υδάτων και θα πρέπει να περιμένουμε 30 εκατομμύρια κόσμος να μετακινηθεί και να μεταναστεύσει. Πού να μεταναστεύσει. Λοιπόν, αυτά τα θέματα έχουν μεγάλη σημασία και συνδέουν την ανάπτυξη με τη μετανάστευση, με το κλίμα, κάτι το οποίο για μας είναι ζωτικό. Θα ακούσουμε λοιπόν τους εμπειρογνώμονες από οργανώσεις των πολιτών, μη κυβερνητικέ οργανώσεις, για να δούμε ακριβώς πώς θα προχωρήσουν τα πράγματα. Έχουμε επίσης ε, προσκαλέσει τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για ε, τους μετανάστες ε, και θέματα εξορίας. Θα ήθελα να δώσω το λόγο λοιπόν πρώτα στην κυρία Πλατόνοβα, η οποία είναι εμπειρογνώμων στο IOM για έξι λεπτά. Η κυρία Πλατόνοβα έχει το λόγο. Λέγομαι Άννα Πλατόνοβα Εκπροσωπώ το Περιφερειακό Γραφείο της Διεθνούς Οργάνωσης για τη Μετανάστευση στις Βρυξέλλες. Είμαστε μια παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση για θέματα μετανάστευσης. Θα ήθελα να θέσω αρκετά θέματα σε αυτή την παρουσίαση σήμερα. Πρώτον, να πούμε τι εννοούμε εμείς όταν ζητάμε συνοχή για την ανάπτυξη, στην πολιτική για την ανάπτυξη και πώς συνδέεται αυτό με το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και τι θεσμικό πλαίσιο θα μπορούσε να συνοδεύει τις τάσεις αυτές. Σε επίπεδο λοιπόν συνοχής των πολιτικών μας, πάρα πολύ συχνά ακούμε για τη συνοχή ανάμεσα στα διάφορα εξωτερικά μέσα και τις εξωτερικές πολιτικές συνοχή ανάμεσα σαν παράδειγμα στην πολιτική στον τομέα του εμπορίου και στην πολιτική στον τομέα της ανάπτυξης. Οι εσωτερικές πολιτικές όμως και αυτές πάρα πολύ συχνά μπορούν να παίξουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της επιρροής του αναπτυξιακού δυναμικού τρίτων χωρών. Αυτό που είναι επίσης σημαντικό είναι η δυνατότητα να βοηθήσουμε στην ανάπτυξη των μεταναστών που κατοικούν στο εσωτερικό της Ένωσης. Τίθενται θέματα εδώ όπως διακρίσεις, ενσωμάτωση του πληθυσμού, όλα αυτά έχουν μεγάλη σημασία. Να αντιμετωπιστούν θέματα όπως η φυγή των εγκεφάλων από φτωχέ χώρες, η σωστή κατανομή δημοσιονομικών πόρων, έτσι ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν αν το αποφασίσουν τις χώρες τους οι μετανάστες αυτοί και σε επίπεδο περιβαλλοντικό και γενικά η παρέμβασή μας παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των τρίτων χωρών. Όταν μιλάμε για πιο συγκεκριμένα θέματα στο εσωτερικό της μετανάστευσης και σχετικά με τους πυλώνες τους οποίους ήδη αναφερθήκατε, όλοι είναι αλληλοσυνδεδεμένοι. Βλέπουμε ποιοι είναι οι κίνδυνοι από τη μετανάστευση, βλέπουμε ποιοι είναι οι σύνδεσμοι της μετανάστευσης με άλλες πολιτικές, η συμπληρωματικότητα της πολιτικής αυτής με άλλες πολιτικές όπως η δημοσιονομική. Όταν μιλάμε για την παράνομη μετανάστευση δεν θα πρέπει να βλέπουμε μόνο τα ad hoc μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού, αλλά θα πρέπει να αναζητούμε και τον τρόπο με τον οποίο οι πολιτικές των αγορών εργασίας μας αυξάνουν ή μειώνουν τη ζήτηση για τέτοιου είδους ε, παράνομες μορφές μετανάστευσης. Όταν συζητάμε θέματα κυκλικής μετανάστευσης θα πρέπει να δούμε αν οι κανόνες μας για την αποδοχή και την εγκατάσταση των μεταναστών τους επιτρέπουν να κυκλοφορούν ελεύθερα και να συνδέονται και με τις χώρες προέλευσης ή είναι αποκλεισμένοι στις χώρες ε, στόχου και ε, φοβούνται να πάνε στη χώρα τους γιατί θα χάσουν τα δικαιώματα διαμονής τους. Το νέο πολιετές τώρα χρηματοδοτικό δημοσιονομικό μάλλον πλαίσιο υπάρχουν προκλήσεις για τη συνοχή εκεί. Είναι σαφές ότι υπάρχει μια επικάλυψη ανάμεσα στις προτεραιότητες εθνικής χρηματοδότησης, ιδιαίτερα όπως το βλέπουν οι δύο γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής που ασχολούνται με τα θέματα. Οι προτεραιότητες των θεματολογικών προγραμμάτων της ΤΕΦΚΟ ε, έχουν σαν στόχο τη διαχείριση των μεταναστών και να συνδέουν τη διαχείριση των μεταναστικών ρευμάτων με θέματα αναπτυξιακά. Όλα αυτά τα θέματα συνδέονται άμεσα με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν να βρούμε τους σωστούς τρόπους χρηματοδότησης και να εντοπίσουμε τρεις τομείς οι οποίοι όπως είπαμε ανησυχούν. Καταρχάς οι επικαλύψεις πρέπει να αποφευχθούν. Ό,τι συνδέεται αυστηρά με την ανάπτυξη δεν θα πρέπει να εμπλέκεται στα θέματα της μετανάστευσης. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ένα παράδειγμα ενός ταμείου σαν παράδειγμα, το οποίο θεωρείται αυστηρά εσωτερικό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ολοκλήρωσης. Λέγει ότι έχει σαν προτεραιότητα την ενσωμάτωση ε, των μεταναστών όταν παλινοστούν στις χώρες προέλευσης. Δηλαδή υπάρχει μια εξωτερική ε, διάσταση σε ένα ταμείο το οποίο είναι αυστηρά εσωτερικό. Τίθεται επίσης και το θέμα της γεωγραφικής επικάλυψης. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι περιφέρειες και οι περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζονται από τα περιφερειακά ταμεία και αν υπάρχουν δύο μέσα χρηματοδοτικά στην ίδια χώρα που ασχολούνται με συγκεκριμένα ταμεία, το θέμα είναι να βρούμε τη σωστή μορφή συντονισμού. Γι' αυτό δημιουργούνται οι λεγόμενες εταιρικές ε, μορφές συνεργασίας, Βλέπουμε ότι και με άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία είναι χώρες που μπορούν να θεωρηθούν χώρες προτεραιότητας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της μετανάστευσης. Γενικότερα προσπαθούμε να δούμε πώς η χρηματοδότηση θα μοιραστεί ανάμεσα στα διαφορετικά μέσα παρέμβασης που υπάρχουν. Έχει ήδη υποθεί από διάφορους εμπλεκομένους, εταίρους κτλ. ότι πρόσφατα κάποια μέτρα, όπως ο πολιτικός διάλογος για τη μετανάστευση, θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από άλλα μέσα ε, και όχι από αυτά τα οποία περιλαμβάνονται στις προτάσεις που ακολουθούμε μέχρι τώρα. Υπάρχουν επίσης ε, και κενά στη χρηματοδότηση της συνεργασίας σε επίπεδο νότου-νότου στον τομέα της μετανάστευσης, σε περιφερειακό επίπεδο, και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ξεκάθαρος ρόλος για τη Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ, η οποία θα πρέπει να παίξει ένα ηγετικό ρόλο. Υπάρχουν και θέματα συμβατότητας σχετικά με το χρονισμό της παρέμβασης και εδώ <clears throat> τα λεγόμενα eco funds και τα αναπτυξιακά ταμεία ε, σε, θεωρητικά ακολουθούν το ένα το άλλο. Δηλαδή από τη μία τα χρήματα του eco και αμέσως μετά έρχονται τα χρήματα της ανάπτυξης. Πρέπει λοιπόν στον χρόνο να υπάρξει σωστή συνεννόηση και συντονισμό. Σε σχέση με τα χρήματα που δίδει το ΕΚΟ υπάρχει το θέμα της δυνητικής επικάλυψης με τα ταμεία άμεσης απόκρισης τα οποία έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένας άλλος τομέας ο οποίος θα πρέπει να εξεταστεί είναι το πώς θα αναγνωρίσουμε θέματα μετανάστευσης σε άλλα εξωτερικά μέσα τα οποία υπάρχουν, κάτι που δεν γίνεται σήμερα. Σαν παράδειγμα το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Αυτές οι εταιρικέ σχέσεις, οι οποίες θα κληθούν να καλύψουν και σχέσεις με χώρες όπως η Βραζιλία, η Κίνα και η Ινδία, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και σαν μέσο για τη βελτίωση του διαλόγου για τη μετανάστευση στα πλαίσια της, του γενικού πολιτικού διαλόγου που έχουμε με τις χώρες αυτές. Ε, άλλοι ομιλητές ε, θα αναφερθούν σε άλλα θέματα και ιδιαίτερα στην ανάγκη για μια σωστή εξισορρόπηση των προτεραιοτήτων χρηματοδότησης στους πυλώνες αυτούς και σε σχέση με συγκεκριμένα έγγραφα και στόχους όπως η στρατηγική 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν μιλάμε για θέματα συνεκτικότητας θα πρέπει να βρούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η ανάπτυξη μιας ευέλικτης πολιτικής μετανάστευσης ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς κάθε φορά και ε, τον σεβασμό φυσικά των δικαιωμάτων των μεταναστών. Υπό το φως όλων αυτών τα οποία προείπα θα πρέπει να δούμε ποιο είναι το σωστό θεσμικό πλαίσιο το οποίο συνοδεύει τον προγραμματισμό και την εφαρμογή αυτών των χρηματοδοτικών μέσων. Και να δούμε και ποιον ρόλο μπορεί να έχουν άλλες γενικές διευθύνσεις στα πλαίσια των διαβουλεύσεων γύρω από τα θέματα αυτά. Και αναφέρομαι εδώ στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, στη Γενική Διεύθυνση Παιδείας, εκπαίδευση συγγνώμη, στον ρόλο της ε, Γενικής ε, ε, Διεύθυνσης Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως επίσης και να μην ξεχνάμε τον ρόλο τον οποίο μπορούν να παίξουν οι αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε μια εσωτερική ομάδα εργασίας η οποία να αντιμετωπίσει όλα τα θέματα συμβατότητας και συνοχής ανάμεσα στα χρηματοδοτικά μέσα εσωτερικά και εξωτερικά που έχει στη διάθεσή της η Ένωση. Δεν θα μακρηγορήσω. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις για όσους ε, για αυτά τα σχόλια τα οποία απευθύνονται στην ε, επικάλυψη που υπάρχει στην ε, δίκησή μας σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και χρηματοδότησης θα παρακαλέσω τώρα την κυρία Μπλοντά Μπουνιό που είναι συντονιστής του προγράμματος Concord να αναφερθεί σε θέματα οι οικογενείες που θεωρεί ότι είναι πολύ σημαντικά για τον χώρο αυτό για, τους, για τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας, λέγομαι Μπλοντίν Μπουνιόν και ε, εργάζομαι εις ε, τις Βρυξέλλες. Ξέρετε ότι το Concord είναι ε, η εξέλιξη της συνεργασίας των μη κυβερνητικών οργανώσεων και μας ζήτησαν να να ε, ε, καταρτήσουμε ε, μία έκθεση σχετικά με την κινητικότητα, τη μετανάστευση, με τα αρχικά ΓΑΜ που θα υποβληθεί το Νοέμβριο. Το ΓΑΜ είναι μία σημαντική πολιτική και αναφέρεται στην πολιτική μετανάστευση η οποία θα διαμορφωθεί στα επόμενα έτη και το Κοινοβούλιο δεν έχει γνωμοδοτήσει τροφοδοτήσει επί του θέματος και πιστεύουμε ότι οι πολιτικές αυτές πρέπει να διατυπώνονται ε, πριν από τη χρηματοδότηση και η χρηματοδότηση πρέπει να υλοποιεί τις πολιτικής. Ακόμη και τώρα με τα χαρά θα αναμείνουμε τα σχόλιά σας αλλά καλό θα ήταν να είχαμε πρώτα την ε, πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα προγράμματα αυτά. Όσο αναφορά την ανάλυση και την δήλωση η οποία έχει καταρτιστεί σχετικά με αυτή την πολιτική δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες αλλά μόνο σε μερικά στοιχεία. Καταρχήν χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ε, παραμένει η ανάπτυξη ένας από τους τέσσερις πυλώνες του προγράμματος αυτού αλλά εντοπίσαμε ε, και κοινά και γι' αυτό έχουμε διατυπώσει οχτώ συστάσεις για να βελτιωθεί το πρόγραμμα αυτό. Καταρχήν ε, ε, εξετάζουμε τα θέματα που ε, άπτονται των μετακινήσεων των πληθυσμών και το, από την άλλη πλευρά ε, με τα θέματα της πολιτικής. Πρέπει να σημειώσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι πρέπει να προωθηθούν τα θέματα αυτά και στους τέσσερις πυλώνες του προγράμματος για του μετανάστες εντοπιζόμενοι και εστιαζόμενοι εις ε, την ε, σωματεμπορία γυναικών και παιδιών. Και ε, θα πρέπει να υπάρξει ισότητα των ε, φίλων που να ε, τονίζεται και σε όλες τις πολιτικές αυτές ε, και στην διατύπωση αποφάσεων. Εδώ μπορεί να παρέμβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να διευκρινίσει αυτό το θέμα. Ε, όσον αφορά την αναπταξιακή πολιτική. Ε, πρέπει να υπάρχει συνέπεια στην πολιτική ε, και συμφωνούμε, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και πολιτική συνεκτικότηση στην ανάπτυξη σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας, διότι τουλάχιστον το πρόγραμμα αυτό δεν πρέπει να εμποδίζει να υλοποιηθούν οι στόχοι και οι συνεργίες θα πρέπει να ισχύσουν για τους τέσσερις πυλώνες για να υπάρξει ε, μία προώθηση όλων των στόχων, πράγμα που αυτή τη στιγμή δεν είναι τόσο προφανές στη διατύπωση των προγραμμάτων. Χρειάζεται μία πολιτική μετακινήσεων που θα εξασφαλίσει ότι η μετακίνηση αυτή θα είναι ασφαλής εναλλακτική λύση για όλους τους εμπλεκομένους και ότι η ανάπτυξη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτών των πολιτικών Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει ένα καλό σύστημα εποπτείας και παρακολούθησης που θα αξιολογεί την πρόοδο των μεταναστών και ε, θα επιτρέψει ε, να υπάρξουν ορισμένες βελτιώσεις ε, συγκεκριμένων πτυχών κατά τρόπον ώστε να συνάδουν οι πολιτικοί πολιτικές αυτές με τους στόχους που έχουν καταρτιστεί. Όσον αφορά τα ε, χρηματοοικονομικά μέσα και την κατανομή ε, των πόρων μεταξύ ταμείων είναι ακόμη ένα θέμα που θα πρέπει να εξετάσουμε διότι υπάρχει μία συνεχής ανησυχητική εξέλιξη ε, δηλαδή υπάρχει μία προσπάθεια ελέγχου των μεταναστευτικών και όλο και περισσότερη βοήθεια δίδεται κατά προτεραιότητα στις χώρες που έχουν μεγάλες μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη για να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα σύνορά τους και ε, αντιθέτως ε, θα πρέπει ε, να υπάρξει μία σαφής καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης για να δοθεί αναπτυξιακή βοήθεια. Για να μπορέσει λοιπόν να προωθήσει κανείς την, τα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανάπτυξη δεν θα πρέπει πρέπει να συνδυάζουμε με προϋποθέσεις την ενίσχυση ε, και με ορισμένες υποχρεώσεις. Θα πρέπει να είμαστε συνεκτικοί με τους στόχους που έχουμε καθορίσει και όχι οι στόχοι να είναι συνεπείς με ό,τι εμείς θέλουμε να κάνουμε και αυτό θα πρέπει να επαναξεταχθεί στο θέμα της χρηματοοικονομικής ενίσχυσης ε, για την μετανάστευση από την Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κανονισμός της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ ε, σχετικά με τα δημόσια αγαθά και τις προκλήσεις η οποία αναφέρεται εις ε, την αντιμετώπιση των προκλήσεων και ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία μικρή αύξηση της χρηματοδότησης για την μετανάστευση και το άσυλο. Αλλά αυτό καλύπτει μόνο δύο από τα τέσσερα προγράμματα τα οποία όπως μας είπε ο συνάδελφός μας αποβλέπουν η καλύτερη ουσιαστικά διαχείριση της μετανάστευσης θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την χορήγηση αναπτυξιακής βοήθειας διότι ε, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε και ζητούμε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξασφαλίσουν ότι ε, θα, ε, θα παρακολουθεί τα θέματα της μετανάστευσης και τώρα θα αναφερθούμε στο ταμείο το οποίο διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων για να στηρίξει ενέργειες ε, που έχουν σχέση με τρίτες χώρες. Δεν σκοπεύουμε ε, να στηρίξουμε ε, δράσεις σε άλλους τομείς ε, και η εξωτερική διάσταση των ε, δύο ταμείων του IMF και του ISF ε, πρέπει να προωθηθεί αλλά να υπάρχει μία συνολική αντιμετώπιση <clears throat> των θεμάτων αυτών διότι η, Τράπεζα Αναπτύξεως και Συνεργασίας επίσης κινητοποιείται σε αυτόν τον τομέα αλλά αυτό δεν προβλέπεται στο σχέδιο του κανονισμού και οι κανονισμοί που αναφέρονται στα ταμεία IMF και ISF δείχνουν ότι υπάρχει η δυνατότητα προωθήσεως των θεμάτων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως χωρίς όμως να συνδυάζονται με τους αναπτυξιακούς στόχους που είναι επίσης προσυμφέρον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε ε, συμπληρωματικότητα ε, μεταξύ των διαφόρων χρηματοδοτήσεων κατά τρόπον ώστε οι πολιτικές που καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Γενικών Υποθέσεων και Εσωτερικών Υποθέσεων να προωθούν τα δικαιώματα των μεταναστών και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και στις χώρες τους προελεύσεως και κατά τη διάρκεια της διελεύσεώς τους από άλλες χώρες και όλα αυτά θα πρέπει να θεσπιστούν στους διάφορους κανονισμούς κατά τρόπον ώστε να μπορέσουν να συνεργαστούν καλύτερα τα διάφορα ταμεία διότι τώρα θα πρέπει να εξασφαλίσουμε επίσης ότι και οι γνωμοδοτήσεις των διαφόρων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα οδεύσουν προς την ίδια κατεύθυνση και σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ε, ήταν μια πολύ καλή παρουσίαση. Δεν ξέρω αν αυτές είναι οι δικές σας απόψεις ή οι απόψεις του προγράμματος Concord και δεν ξέρω ε, ε, αν αντιμετωπίζουν τα ερωτήματα τα οποία έχουμε θέσει και που αναφέρονται εις τα συμφέροντα του Ευρωπαίου φορολογουμένου. Μας είπατε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και δύο γιατί θα πρέπει να αναπτυχθεί μία πολιτική καταρχήν και ε, όταν υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες και πολλοί άνεργοι στην Ευρώπη ε, θα πρέπει να σκεφτεί κανείς και τους γυρεότερους Ευρωπαίους δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει στο πρόγραμμα κάτι για όλους και για τους φτωχούς και για τους πλουσίους και παρακαλώ τώρα την κυρία Ντοπολού. Ναι. Το λόγο έχει η κυρία Παπαδοπούλου. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προσφύγων, ε, μια ε, συνεργασία 70 μη κυβερνητικών οργανισμών από χώρε όπω η Πορτογαλία, ή το Αζερμπαϊτζάν, πολλέ μη κυβερνητικέ οργανώσει επίση που δραστηριοποιούνται σε τρίτε χώρε και παρέχουν βοήθεια σε προσφύγε και εκτοπιστέτε ε, ανά τον κόσμο. Είμαστε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει ανάγκη να τονίσουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την προστασία των προσφύγων και τη συζήτηση για τους μηχανισμούς βοήθειας. Είναι σημαντικός ο μηχανισμός DCI και πρέπει στο πλαίσιο αυτό να θέσουμε κάποια ζητήματα. Τρία βασικά πράγματα θα σχολιάσω. Πρώτα απ' όλα προστασία προσφύγων και πώς εντάσσεται ε, ε, στην ανακοίνωση για την κινητικότητα καθώς επίσης και πρόταση για DCI και ε, θεματικό πρόγραμμα. Ποιε είναι οι προκλήσει, επίση η σχέση μεταξύ των μηχανισμών εξωτερική βοήθεια ε, και με το μηχανισμό ε, για του πρόσφυγε, πώ αλληλοσυνδέονται, αν αλληλοεπικαλύπτονται και πώ. Και τρίτο θέμα, ρόλο και συμμετοχή οργανισμών τη κοινωνία των πολιτών στα δύο είδη χρηματοδότηση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, Έχουμε κάποια σχόλια πρόσφατα δημοσίευση σε σχέση με αυτήν την ανακοίνωση για να δούμε ακριβώς πού εντάσσεται σε αυτήν ε, τη στρατηγική προστασία των προσφύγων. Το βασικό μας σχόλιο είναι ότι η συνολική προσέγγιση στην κινητικότητα και τη μετανάστευση είναι ένα πλαίσιο που κατά κύριο λόγο επικεντρώνεται στη διαχείριση της μετανάστευσης και πλέον όλο και περισσότερο στην κινητικότητα. Η προστασία των προσφύγων είναι ευπρόσδεκτο ως ε, στοιχείο για καλύτερο συντονισμό, αλλά πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει πιο θαραλέα στάση και να παρουσιάσει μια πληρέστη, μια συνεκτικότερη πολιτική και για τη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες και τους εκτοπιστέντες, υπερβαίνοντας το στρενό όριο της μετανάστευσης. Βλέπουμε τι γίνεται με διάφορα μέσα και μηχανισμούς που είναι προγράμματα της ανθρωπιστικής βοήθειας από τα οποία αποφελούνται ε, οι πρόσφυγες. Αλλά βλέπουμε να μην υπάρχει συνεκτικότητα, να μην υπάρχει συνέπεια και ξεκάθαρη στόχη ε, στρατηγικής και πολιτικής σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες. Θα θέλαμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλάβει τη θέση που τη αρμόζει στο διεθνέ προσκήνιο και να καταστεί ένα πρωταγωνιστής ε, σε παγκόσμιο επίπεδο στο θέμα τη προστασία των προσφύγων. Και αυτό έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο τα χρηματοδοτικά μέσα λαμβάνουν υπόψη τους ε, ζητήματα των προσφύγων δεν είναι ε, θέμα επαρκούς χρηματοδότησης, γιατί η χρηματοδότηση υπάρχει και υπάρχουν προγράμματα εδώ και χρόνια τα οποία στηρίζουν αυτούς τους πληθυσμούς. Το θέμα είναι αν γίνονται συνεπείς και συνεκτικές προσπάθειες για την προώθηση λύσεων ε, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, διότι δεν πρόκειται για μια μεμονωμένη κοινότητα. Μιλάμε για εκατομμύρια άτομα, ε, πρόσφυγες δηλαδή, που πρέπει να τύχουν προστασίας. Αν δούμε τώρα το θεματικό πρόγραμμα του Challenges και τη σχέση με το άσυλο και την μετανάστευση, πρέπει να πω ότι υπάρχει αναφορά σε κάποιες περιφερειακές και εθνικές πολιτικές ε, για το άσυλο. Αλλά θεωρούμε ότι περιορίζονται οι προσπάθειες στη διαχείριση της μετανάστευσης. Θα θέλαμε η προστασία των προσφύγων και η παροχή βοηθείας να ε, είναι πιο συγκεκριμένο στόχο στα διάφορα προγράμματα. Παραδείγματο χάρη, η προστασία, η βοήθεια των προσφύγων θα πρέπει να ενταχθεί στο Ευρωπαϊκό Μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίσης, να περιλαμβάνεται αυτή η διάσταση στα διάφορα γεωγραφικά μέσα και εργαλεία. Με στόχο μια μεγαλύτερη συνεκτικότητα και μια πιο τολμηρή πολιτική προστασία των προσφύγων. Σε ό,τι αφορά τη σχέση μεταξύ των δύο ειδών ε, μέσων, τα εξωτερικά και τα εσωτερικά, υπάρχει κίνδυνος αλληλεπικάλυψης μεταξύ της εξωτερικής διάστασης ε, και των εξωτερικών μηχανισμών βοήθειας. Τι χρηματοδοτείται από ποιο μηχανισμό. Προγράμματα περιφερειακά, παραδείγματος χάρη, ε, επιστροφή και επανένταξη των προσφύγων. Πού χαράσουμε διαχωριστικέ ε, γραμμέ, τι είναι δημιουργία ικανοτήτων, capacity building για πρόσφυγε, τι δεν είναι, τι καλύπτεται ε, στα περιφερειακά προγράμματα από τα εγχώριου πόρου και τι από την εξωτερική βοήθεια. Η επανεγκατάσταση πού καλύπτεται, πού εντάσσεται κτλ. κτλ. Και δεν είναι ένα θέμα διευκρίνησης απλά και μόνο, είναι και θέμα μερίσιας διάταξης Υπάρχουν ε, εγωκεντρικοί, ε, αν, θέλετε, στόχοι ε, στην, στα εσωτερικά κονδύλια, αλλά τα αναπτυξιακά κονδύλια έχουν διαφορετικά, διαφορετικούς στόχους, δηλαδή θέλουν να προωθήσουν λύσεις σε τοπικό επίπεδο. Και πρέπει να υπάρχει συνεκτικότητα και συνέπεια με τους στόχους. Υπάρχει επίση ανάγκη συνεκτικότητα μεταξύ τη εξωτερική διάσταση ε, στα εγχώρια κονδύλια και στου μηχανισμού εξωτερική βοήθεια. Και θα θέλαμε να υπάρχει μια υποχρεωτική διάταξη ε, στην πρόβλεψη ε, για τα εγχώρια κονδύλια ώστε να υπάρχει αυτή η διασύνδεση με όλες τις δράσεις οι σχετίζονται με την εξωτερική διάσταση. Εξωτερική διάσταση μετανάστευσης και πρόσφυγες, άσυλου. δίνει το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση δυνατότητα στα κράτη-μέλη να ε, κινητοποιηθούν και σε τρίτε χώρε μέσω εθνικών προγραμμάτων. Και αυτό είναι μια καινοτομία, ένα νοτερισμό. αλλά υπάρχουν κίνδυνοι κατά την άποψή μα. Πώ θα εξασφαλίσουμε δηλαδή να είναι συνεπεί οι δράσει αυτέ με την αναπτυξιακή πολιτική και του στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα αυτό στι σχετικέ χώρε και να μην αντικατοπτρίζουν μόνο διμέρη πολιτικά συμφέροντα, ούτε να στρέφονται κατά τη αρχή τη αλληλεγγύη σε σχέσεις με τη συνεργασία μας με τρίτε χώρες. Υπάρχει η κατεπίγουσα βοήθεια, emergency assistance, που προβλέπεται στο Ταμείο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο και εκεί μπορεί να υπάρξει αλληλεπικάλυψη με το μέσο που υπάρχει αυτή τη στιγμή για τη σταθερότητα, διατάξει ειδικών μέτρων στο πλαίσιο του DCI κτλ. Όλα αυτά δυνητικά θα μπορούσαν να ανταποκριθούν στην ανάγκη υπάρξη κατεπίγουσα βοήθεια, αλλά δεν ξέρουμε πώ όλα αυτά μπορεί να είναι συμβατά χωρί να υπάρχουν αλληλεπικαλύψει. Τέλο, σε σχέση με τον ρόλο και τη συμμετοχή τη κοινωνία των πολιτών στα μέσα και μηχανισμού αυτού, τα γεωγραφικά μέσα προβλέπουν τη δυνατότητα διαβούλευσης με τους χρηματοδότες και με τους διεθνούς οργανισμούς αλλά και την ε, ε, τοπική κοινότητα των πολιτών όπου δει. Στην πρόταση για την εξωτερική διάσταση λέγεται shall consult. Διαβουλεύονται, είναι μια ε, υποχρέωση και το επικροτούμε. Θα θέλουμε λοιπόν να συστήσουμε οι οργανώσεις της των πολιτών και οι διεθνείς οργανισμοί να αποτελέσουν τμήμα των συζητήσεων και των διαβλέψεων πριν από τον προγραμματισμό, διότι είναι οι οργανώσει που διαστροπούνται επί τόπου, έχουν ε, καθημερινέ επαφέ με ε, ετούντε άσυλο, με πρόσφυγε, ε, με μετανάστε, ξέρουν, αφουγκράζονται τι ανάγκε και πρέπει να είναι και εκεί για να βλέπουν ότι πραγματικά ο προγραμματισμό αντιστοιχεί στι ανάγκε του πληθυσμού. Ευχαριστώ. Εμεί σα ευχαριστούμε, λέει ο για αυτή την παρουσίαση. Η εντύπωση που έχω αποκομίσει ακούγοντα του τρει εμπειρογνώμονε είναι ότι δεν είναι ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο εμεί συντονίζουμε και του στόχου με τη χρηματοδότηση κτλ. Φίλιπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι ένα πολύ επίκαιρο θέμα πράγματι και δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα με την πρόσωπο της οργάνωσης Concord. Καλύτερα θα ήταν πρώτα να συζητήσουμε για πολιτική και μετά για χρηματοδότηση μέσων. Ωστόσο, νομίζω ότι πρέπει να δούμε το θέμα λίγο πιο βαθιά. Δεν αρκεί η πολιτική. Αλλιώς θα περιοριστούμε στην ε, γνωστή συζήτηση ε, πώς οι μετανάστες μπορούν να εισέλθουν σε μια χώρα, να πάρουν καθέσεις κτλ. Ε, ή στην Ελβετία που υπάρχει και το θέμα από πού προέρχονται ή από πού πρέπει να προέρχονται οι μετανάστες. Το θέμα λοιπόν που προκύπτει είναι ισχύει αυτή βάση ε, first come, first served. Όλοι είμαστε αν θέλετε μετανάστες. Κάποιοι φτάσανε πρώτοι κάπου. Και αυτοί έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν ποιος έχει το δικαίωμα να ενταχθεί σε κάποιο μεταγενέστερο στάδιο. Νομίζω ότι η συζήτηση, ναι είναι επίκαιρη, είναι και δύσκολη όμως, διότι πολλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι μπορούν να υπαγορεύσουν ποιοι είναι οι νόμιμοι μετανάστες και ποιοι όχι. μπορούμε να συζητήσουμε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αλλά όσο υπάρχει αυτή η αρχή και αν μπορούν τα κράτη-μέλη απλά ε, να αποφασίζουν για τη νόμιμη διαμονή παρουσία ενός ατόμου ή τη μη νόμιμη παρουσία του σε ένα κράτος, δεν πρόκειται να λυθούν τα προβλήματα. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν. Μπορούμε να ασκήσουμε πιέσεις σε εκείνα τα κράτη-μέλη για να δουν το ζήτημα και το πρόβλημα της μετανάστευσης με ε, ένα πιο σφαιρικό μάτι, πιο σφαιρικό τρόπο. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα. Δεν ήταν πάντα έτσι τα πράγματα. Υπάρχει αρνητική αντίληψη πλέον για τη μετανάστευση, για τους μετανάστες. Μπορεί να αναστραφεί κάτι τέτοιο και να θεωρηθεί η μετανάστευση κάτι θετικό ευχαριστώ, Φίλιππ, για την ενδιαφέρουσα παρέμβασή σου. Παρακαλώ τον Ρικάρντο να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τις τρεις προσκεκλημένες μας. Ήταν πολύ διαφωτιστικές παρουσιάσεις τους για ένα τόσο σημαντικό και τόσο επίκαιρο ζήτημα. Είμαστε σε μια φάση όπου η μετανάστευση δεν μιλάμε καν μόνο για μετανάστες, μιλάμε και για τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά πιστεύω ότι χάνουμε την γενικότερη εικόνα και πρέπει να κάνουμε και μια ιστορική αναδρομή και να δούμε η Ευρώπη 1860-1870 μέχρι το 1920 πώς ήταν, δεν υπήρξαν πολλοί Ευρωπαίοι που μετανάστευσαν, ε, δεν είναι η Ευρώπη μια ήπειρος ε, με έντονα μεταναστευτικά ρεύματα. Είδαμε και τόσους καταβλισμούς ε, ε, προσφύγων. Και στα Βαλκάνια μέχρι σύντομα, μέχρι πρόσφατα μάλλον. Άρα πρέπει να σκεφτούμε και να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό ότι ε, μην ξεχνάμε ότι κάποτε μεταναστεύσαμε κι εμείς. Το αντίθετο έχει σχέση. Είμαστε η Ήπειρος ε, με τα μεγαλύτερα ποσοστά μετανάστευσης προς άλλες χώρες και τώρα είμαστε μια Ήπρος που υποδέχεται μετανάστες. Πώς μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε. Πώς θα συνδυάσουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Πρέπει να το σκεφτούμε λοιπόν στο πλαίσιο του μελλοντικού, έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, σταθερότητα ε, των ομάδων επίσης. Δημιουργία σταθερών ομάδων ε, σε σχέση με την μετανάστευση. Είναι ένα σημαντικό θέμα στην Ευρωλατινοαμερικανική συνέλευση υπάρχει αυτή η σταθερή ομάδα, για παράδειγμα. Υπάρχουν βουλευτές από τη Λατινική Αμερική και βουλευτές από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι οποίοι καταφέρνουν να ε, καταλήξουν σε συμφωνίες σε θέματα μετανάστευσης και έτσι προκύπτουν κοινέ θέσει, ε, τι οποίε μπορούν να δεχτούν οι περισσότεροι βουλευτέ. Θα μπορούσαμε προ αυτή την κατεύθυνση να κινηθούμε ακόμη περισσότερο, αυτό το σχηματισμό κάποιων σταθερών ομάδων θα συζητήσουμε και για τον DCI και τον όλο προβληματισμό για τα κονδύλια αυτού του μέσου, αν θα φτάσουν στην καταπολέμηση της στόχης και τα λοιπά, να μην δημιουργηθεί ανασφάλεια. Είναι όλα θέματα τα οποία είναι ενδιαφέροντα και θα τα συζητήσουμε στη συνέχεια. Δυστυχώς, αληθεύει ότι δεν έχουμε ξεκινήσει από το μηδέν. Αντίθετα, έχουμε συναντήσει πολλά προβλήματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Ολοκληρώνοντας, συμφωνώ με την τελευταία ομιλήτρια ότι πράγματι και δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Πρέπει να ακούσουμε ε, την κοινωνία των πολιτών, όλες τι οργανώσεις που εργάζονται επί τόπου και για τη μετανάστευση και για τους πρόσφυγες. Πρέπει να ακούσουμε ε, τι γίνεται επί τόπου ε, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια πολιτική με τα λόγου γνώσεως, έχοντας υπόψη στο τι συμβαίνει επί τόπου. Uh, thank you, Ricardo. May I Augustine to make his comment? Αγκουστίν, παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Σας συγχαίρω που περιλάβατε στην ημερήσια διάταξη της Επιτροπής ΔΕΒ ένα τόσο σημαντικό θέμα. Μία πρώτη σύσταση. Νομίζω ότι θα ήταν ίσως ε, καλύτερο, πιο εμπλουτιστικό, αν θέλετε, να έχουμε μια κοινή συνεδρία τη Επιτροπή ε, Πολιτικών Ελευθεριών και τη Επιτροπή Ανάπτυξη για να συζητήσουμε από κοινού το θέμα αυτό. Για ποιο λόγο, διότι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχει μακρά εμπειρία στον τομέα της μετανάστευσης και έχει κάποιο προκαθορισμένο δόγμα, αν θέλετε. Δηλαδή, ε, στην Επιτροπή Ελευθεριών ποτέ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο όρος παράνομος, illegal, ε, για, κάποιες, ε, για μετανάστες. Χρησιμοποιούμε τη λέξη ε, irregular και όχι illegal. Αυτός δηλαδή που δεν έχει τακτοποιήσει υποχρεώσεις τους, που δεν έχει τα επίσημα έγγραφα. Και έχουμε όλα αυτά τα θέματα, την ένταξη, τη διεθνή η επικουρική προστασία, την επιστροφή, την ανάπτυξη, τους πρόσφυγες κτλ. Εδώ όπως θα θυμάστε κύριε Πρόεδρε και παρουσία της κυρίας Άστον, είχαμε ε, καταγγείλει το ότι δεν είναι καθόλου σωστό ε, τα αναπτυξιακά ε, κονδύλια να είναι αυτά τα οποία ανέφερε και η κυρία και να το συνδέουμε με τον έλεγχο των συνόρων. Διότι αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον κοινωνού. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε να πηγαίνουν αυτά τα χρήματα στην προστασία, στον έλεγχο των συνόρων. Υπάρχουν τέσσερα ειδικά ταμεία την άλλη πλευρά. Εσείς χρηματοοικονομικές, στις δημοσιονομικές μάλλον προοπτικές που θα εγκριθούν. Είναι τα τέσσερα ταμεία, ένα από αυτά είναι για τους πρόσφυγες, για το άσυλο άλλο ένα και για τον έκτο εξωτερικών συνόρων ε, και το για τη μετανάστευση. Επομένως, τέσσερα ταμεία με πολύ ξεκάθαρες ε, αρμοδιότητες και δεν θα πρέπει να τα συγχαίουμε με τα ειδικά ταμεία για την ανάπτυξη ή για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ολοκληρώνοντας, το σχόλιο μου, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω κάτι το οποίο έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη περιοχή του κόσμου, που θα τη συζητήσουμε απόψε και θα ψηφίσουμε μάλιστα, Λατινική Αμερική. Λατινική Αμερική για ανάπτυξη. Πρέπει να γνωρίζετε ότι στο Αμβούργο την επόμενη εβδομάδα ε, θα συνεδριάσει η Eurolat, η οποία θα συζητήσει μεταξύ άλλων ένα πολύ σημαντικό ζήτημα που νομίζω ότι ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή Ανάπτυξης θα πούμε στην κυρία Φερέρο Βάλτνερ, στην Πενίτα Φερέρο Βάλτνερ, την επίτροπό μα, που είναι πρόεδρος του ιδρύματο για Ευρωπαϊκή, Λατινική Αμερική και Καραϊβική. Θα τη πούμε λοιπόν ότι με προσωπική δέσμευση του Προέδρου του Κοινοβουλίου θα δημιουργηθεί ένα παρατηρητήριο για τη μετανάστευση. Για ποιο λόγο? Για να έχουμε την επιστημονική και πολύ πιο συγκεκριμένη αντίληψη του τι συμβαίνει με το μεταναστευτικό φαινόμενο ένθεν κακήθεν. Σε και σε αυτή την περιοχή και ε, στην, ε, στη δική μας περιοχή και στη Λατινική Αμερική. Θα ήθελα λοιπόν ε, η Επιτροπή Ανάπτυξης να συμμετάσχει σε αυτή την πρωτοβουλία γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε πολύ συγκεκριμένα πώς αναπτύσσεται το φαινόμενο της μετανάστευσης ένθεκα και του Ατλαντικού. Αυτά είχα να πω και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Uh, ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Η ιδέα για την κοινή συνεδρίαση ανάμεσα στην Επιτροπή Ανάπτυξης και τις Δημόσιες Ελευθερίες είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί σε επίπεδο συντονιστών. Και η Γραμματεία θα το φροντίσει. Σας ευχαριστώ για την πρόταση. Η συζήτηση αυτή πράγματι παρουσιάζει ιδιαίτερα ενδιαφέρον και εννοώ τη συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. I think it is not just the case that... Uh, Νομίζω ότι Πολλοί από τους προηγούμενους ομιλητές μας θύμισαν ότι όλοι είμαστε μετανάστες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας σε αυτήν εδώ την αίθουσα που να μην έχει γονείς, συγγενείς ή προγόνους γενικά οι οποίοι να μην έχουν μεταναστεύσει εδώ και εκεί. Θα πρέπει λοιπόν το θέμα της μετανάστευσης να το αντιμετωπίσουμε με πολύ ανοιχτή διάθεση. να τολμήσουμε να μιλήσουμε ειλικρινά για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ελέγξουμε ε, τις ροές τις μεταναστευτικές χωρίς να αγνοούμε σε καμία περίπτωση το πολιτιστικό κομμάτι αυτού του φαινομένου, χωρίς να αγνοούμε το ποιοι είμαστε εμείς, το πώς φτάσαμε εδώ, το από πού ήρθαμε και νομίζω ότι αν δεν τα αγνοούμε όλα αυτά, οι λύσεις που θα δώσουμε θα είναι καλύτερες και οι προοπτικές για τις νέες γενιές πιο ελπιδοφόρες. Χαίρομαι λοιπόν που ακούσαμε τους εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών. Οι παρεμβάσεις τους τελικά ήταν ενθαρρυντικές. Ελπίζω και εμείς με τη σειρά μας να μπορέσουμε να τους ενθαρρύνουμε για να εργαστούν σε αυτόν τον πολύ ευαίσθητο χώρο. Οι προσπάθειες που κάνουν οι ΜΚΟ είναι τεράστιες. Θα πρέπει να αξιολογηθούν πολύ περισσότερο από όσο εκτιμώνται σήμερα. Το θέμα δεν είναι η συνεισφορά σας σε αριθμητικό ή επίπεδο ποσοστών στην ανάπτυξη των χωρών αυτών κτλ. και στο πόσο ελέγχεται ή δεν ελέγχεται ή επηρεάζεται τον έλεγχο της μετανάστευσης. Να υπογραμμίσω ένα επιπλέον σημείο. Είναι θετικό να υπάρξει μια πρωτοβουλία, να υπάρχει μια πρωτοβουλία έτσι ώστε το θέμα της μετανάστευσης και στο δικό μας κοινοβούλιο να το αντιμετωπίσουμε σε επίπεδο πολλαπλών, αν θέλετε, αντιλήψεων. Γιατί πρόκειται για ένα εξαιρετικά πολιτικό θέμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην θελήσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων μερικές φορές. Τα μεταναστευτικά ρεύματα επανειλημμένα είναι συνέπειες κλιματολογικών αλλαγών, άλλων φυσικών θα έλεγα αιτίων, που δεν είναι ανθρωπογενή. Αλλά έχουμε όμως και ανθρωπογενείς μεταναστευτικές ροές και αυτό ε, πρέπει να το αναγνωρίσουμε και είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε τις ανάγκες των μεταναστών από τη μία, τις ανάγκες των ετούντων άσυλο, με το ότι η διεθνής κοινότητα είναι αργή, καθυστερή και δεν λύνει τα προβλήματα. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, δεν είναι φυσιολογικό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε το ότι έχουμε εκατοντάδες χιλιάδες μεταναστών προσφύγων που ζουν σε τέντες για δεκάδες χρόνια. Και θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με, του νέου είδους, με τους νέου είδους μετανάστες. Ε, η νέα γενιά, σαν παράδειγμα στα στρατόπεδα των Παλαιστινίων προσφύγων, δεν βλέπουν το μέλλον ε, με τις ίδιες προοπτικές και τις ίδιες ανάγκες όπως οι γονείς τους και οι νέοι αυτοί ζουν σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο, έχουν ανάγκη να πάρουν μέρος σε αυτόν τον ε, παγκοσμιοποιημένο κόσμο και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να, να αγνοούμε εμείς. Δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλους τους μετανάστες σαν gastarbeiter και δεν πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλους τους μετανάστες σαν ανθρώπους οι οποίοι απλά προσπαθούν να επιβιώσουν οριακά. Όχι, υπάρχουν πιο περίπλοκες και σύνθετες περιπτώσεις μεταναστευτικών ρευμάτων και φαινομένων σήμερα. Δεν μπορούμε επίσης να αρκεστούμε στο να είμαστε ο ισχυρότερος αν θέλετε σαν Ευρωπαϊκή Ένωση ομιλώ ε, παροχέας βοήθειας στον κόσμο. Θα πρέπει να δώσουμε περισσότερα χρήματα και στην αναπτυξιακή βοήθεια, σε είδη βοηθείας εν πάση περιπτώσει που θα βοηθήσει και αυτούς οι οποίοι ζουν σε στρατόπεδα προσφύγων, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι αναζητούν ένα καλύτερο περιβάλλον προσωπικής εξέλιξης και εργασίας. Οικονομικά εννοώ. Τελειώνοντας να πω ότι το θέμα που έχουμε μπροστά μας θα το συζητάμε για πάρα πάρα πολύ καιρό. Και δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα αυτό μόνον όταν σε ορισμένες χώρες ένα νέο πολιτικό κόμμα, σαν παράδειγμα με κάπως ιδιόρυθμες πολιτικές βλέψεις έρχεται στην εξουσία και δημιουργούνται περαιτέρω, ενισχύονται περαιτέρω τάσεις έλλειψης ανοχής απέναντι στους μετανάστες, απέναντι σε εκπροσώπους διαφορετικών πολιτισμών. Αντίθετα θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το θέμα, το πρόβλημα και ε, θα πρέπει να το συζητάμε περισσότερο, θα πρέπει να το συζητάμε πολύ περισσότερο όχι μόνο στους νέους οι οποίοι πιστεύουν ότι πρέπει να ελαφρύνουν την ανθρώπινη δυστυχία και ασχολούνται με αυτό, αλλά θα πρέπει να ενημερώσουμε σωστότερα όλους ε, τους, ε, όλους τους πολίτες της Ένωσης, γιατί πρόκειται για σοβαρότατο θέμα. Αναφερθήκατε και στις εξωτερικές υποθέσεις. Και Νομίζω ότι υπάρχει εκπρόσωπος ε, της ε, διευθύνση αυτής ε, που θα περάσει το μήνυμά μας. Θέλω τώρα να ζητήσω στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας παρουσιάσει τα σχόλιά της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ωραία. Νομίζω ότι όσον αφορά το βασικό στόχο που είναι ε, ο διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων μέτρων που έχουν προταθεί και έχουμε μία σαφή πολιτική ανάπτυξης. Η μετανάστευση προβλέπεται ή στην πολιτική αλλά και στην Agenda for Change που είναι ε, το πολιτικό πλαίσιο για τις δράσεις μας ε, για το δημοσιονομικό μέτρο επαριθμών 4 και λέγεται ότι πρέπει ε, να προωθήσουμε τις πολιτικές που διευκολύνουν διευκολύνουν την περιφερειακή κινητικότητα εργασίας και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βοηθήσει τις υποανάπτυξη χώρες να ενισχύσουν τις πολιτικές τους και τις δραστηριότητες τους στη μετανάστευση και την κινητικότητα για να αυξηθεί η επίπτωση της ανάπτυξης σε αυτά τα πλαίσια. Δηλαδή τα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει, όποια και να είναι, είτε είναι θεματικά είτε γεωγραφικά, θα έχουν σαν στόχο να προωθήσουν αυτό το δεσμό της μετακίνησης και της ανάπτυξης προς όφελος των συνεργαζομένων χωρών και των μεταναστών. Και νομίζω ότι έτσι υπάρχει μία συνεκτική προώθηση ε, της Agenda for Change με τις ε, GAMP. Ε, πράγμα το οποίο έχουμε διατυπώσει στους τέσσερις στόχους που καταρτίστηκαν για τα θεματικά προγράμματα. Όταν μιλάμε λοιπόν για τη διακυβέρνηση της μετακίνησης εννοούμε ότι πρέπει κανείς να εξετάσει πέραν των ποσοτικών κριτηρίων και τα θέματα διακυβέρνησης γιατί πολλές χώρες δεν έχουν υπολογίσει το βάρος ε, της μετανάστευσης ε, ε, στην οικονομία είτε γιατί είναι χώρες εξαγωγικές μετανάστευσης ή γιατί δεν έχουν υπολογίσει παραδείγματος χάρη όπως η Λιβύη ή η ακτή του ελεφαντοστού ότι την επίπτωση της μειώσεως του εργατικού δυναμικού στη γεωργία και θα πρέπει και οι χώρες αυτές να καταλάβουν καλύτερα και να εννοήσουν την σημασία της μετανάστευσης στην δικιά τους ανάπτυξη. Οπότε όσον αφορά το διαχωρισμό των διαφόρων μέτρων, νομίζω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος, μπορεί να ε, υπάρξει μία τέτοια έννοια, αλλά πρέπει να δούμε πώς ε, καταρτίζουμε τα κριτήρια επιλεξιμότητος και είναι σαφές ότι πρόκειται για μέτρα εξωτερικής βοηθείας που αποτελούν μια βασική πηγή χρηματοδότησης όσον αφορά τη χρηματοδότηση με τις τρίτες χώρες. Και υπάρχουν βέβαια και συγκεκριμένοι στόχοι, αλλά το μέτρο αυτό δεν θα επικαλύπτεται, αλλά μάλλον θα συμπληρώνει τις, ε, τα μέτρα προτεραιότητας για την αναπτυξιακή ε, συνεργασία και η λογική μας είναι να υπάρχει εδαφική συνέχεια, δηλαδή να υπάρξουν δράσεις που ξεκινούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά πρέπει να συνεχιστούν ή στις χώρες υποδοχής. Παραδείγματος χάρη για την υποδοχή της μετανάστευσης ή τις διατυπώσεις πριν από μία νόμιμη μετανάστευση η οποία είναι αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την ε, ε, ε, ε, αναπτυξιακή συνεργασία κοιτάξαμε το θέμα των παρανόμων μεταναστών των εθελοντών και η ε, στήριξη για να μπορέσει να υπάρχει κάποια μετατόπιση και πανεγκατάσταση των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε τέσσερα μέτρα που προωθούμε ε, ε, δράσεις οι οποίες δεν προωθούν μόνο την ανάπτυξη αλλά και τις εσωτερικές ευρωπαϊκές πολιτικές εκτός της ευρωπαϊκής επικράτειας. Υπάρχουν συνεργασίες ιδίως βραχυπρόθεσμες και ενδεχομένω μέσο πρόθεσμες για ορισμένε δράσεις και ιδίω προ όφερο τη ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τις εξωτερικές συνεργασίες και με τις εξωτερικές υπηρεσίες των εμπλεκομένων χωρών ή περιφερειών. Εάν λοιπόν ε, ε, θυμόμαστε αυτό το πλαίσιο και το πλαίσιο πλαίσιο της ε, αναπτυξιακής ε, ε, συνεργασίας δεν θα υπάρχουν επικαλύψεις αλλά αμοιβαίε προωθήσεις όπως στις συνεργασίες κινητικότητος όπου θα υπάρχει συγχρηματοδότηση για διάφορα μέτρα. Σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε εάν μακρηγόρησα ευχαριστώ. Με συγχωρείτε που χρειάστηκε να σας κόψω, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν στις αξιολογήσεις σας έχετε λάβει υπόψη την ε, αξία των ε, καταβολών, δηλαδή ε, των χρημάτων που μπορούν να σταλούν πίσω στις χώρες, δηλαδή για να δείτε ποιες είναι οι επιπτώσεις αυτών των καταβολών συναλλάγματος. Ναι, στην ανάπτυξη ορισμένων χώρων χωρών. Σκέφτηκα το Ταζικιστάν του οποίου 50% εξαρτάται ε, από τις ε, ε, από τις εισαγωγές των μισθών των ξενιτεμένων, 13% για τις Φιλιππίνες, 30% για τη Μολδαβία, αλλά οι Φιλιππίνες παραδείγματος χάρη θεωρούν ότι το κόστος το οποίο υπάρχει για να υπάρχει ε, μία πλαισιωμένη πολιτική μετανάστευσης ε, είναι πολύ υψηλό ε, και αμφισβητούνται ε, τα θετικά αποτελέσματα σε πολλούς τομείς. Θεωρούν ότι το κοινωνικό κόστος είναι πολύ σημαντικό για τις οικογένειες, για τα παιδιά που μένουν πίσω. Τίθενται ερωτήματα και μας ζητούν να ξαναπροσανατολίσουν την οικονομία τους και ε, να αναδιοργανώσουν τις μεταναστεύσεις χωρίς ε, να υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις. Πρόκειται λοιπόν για ουσιαστικά ε, μία σωστή διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και έχετε ένα έγγραφο στην γάμπ στην πολιτική αυτή που προαναφέραμε και εκεί αναφέρονται οι επιπτώσεις ε, των ε, μεταναστευτικών ροών και ιδίως στο οικονομικό βάρος ε, των μεταναστεύσεων για την ανάπτυξη μιας χώρας και αυτά είναι θέματα τα οποία θέλουμε να εμβαθύνουμε με τα μέτρα τα οποία έχουμε προτείνει για τις επόμενες προοπτικές που θέλουμε να καταρτήσουμε. Ευχαριστώ. Όταν θα υπάρξει μία κοινή συνεδρίαση με την μεταξύ Επιτροπής Ανάπτυξης ε, και Οικονομικής Επιτροπής θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε. Υπάρχει κόστος για αυτές τις καταβολές των μισθών από το εξωτερικό. Και αυτό δεν το έχουμε συζητήσει. Ε, Επανέρχομαι λοιπόν στους, στους εμπειρογνώμονες χωρίς χρόνο για συζήτηση γιατί δεν μας περισσεύει. Κάρλος, μία σύντομη παρέμβαση ενός λεπτού. Ευχαριστώ. Είμαι από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Υποθέσεις. Αφού είπατε ότι δεν έχω πολύ χρόνο στη μου, απλά θα επιβεβαιώσω ποια είναι η λογική πίσω από αυτήν ε, τη συνιστός εξωτερικής διάστασης για το μελλοντικό κονδύλιο στο πλαίσιο των εσωτερικών υποθέσεων. Ο στόχος λοιπόν ουσιαστικά δεν είναι η αλληλεπικάλυψη, η επανάληψη όσων ήδη γίνονται με τα μέσα εξωτερικής βοήθειας. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να παράσχουμε μια πιο επαρκή χρηματοδότηση, γιατί τα υφιστάμενα μέσα δεν είναι τα καλύτερα ε, δυνατά για κάποιες από τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Επιτροπή Ανάπτυξης είχαμε και κατά το παρελθόν συζητήσει το θέμα αυτό και νομίζω ότι πολύ σωστά είχε επισημανθεί ότι για να χρησιμοποιηθεί το θεματικό πρόγραμμα για τη στήριξη δράσεων που σχετίζονται με την υλοποίηση συμφωνιών επανεισδοχής δεν ήταν και ό,τι καλύτερο. Γιατί το θεματικό πρόγραμμα δεν έχει αυτό το βασικό τουλάχιστον στόχο. Στις συζητήσεις λοιπόν που είχαν γίνει ε, προτάθηκε αυτή η εξωτερική διάσταση η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δράσεις και τα μέσα που θα χρηματοδοτηθούν θα είναι κάποια μέσα που σχετίζονται με τις συμφωνίες περί επανεισδοχής. Υπάρχει το πρόβλημα της αλληλεπικάλυψης. Προσπαθήσαμε και καταφέραμε νομίζω να βρούμε μια διαχωριστική γραμμή. Άρα έχουμε και τους μηχανισμούς συντονισμού είτε σε επίπεδο Βρυξελών είτε και σε επίπεδο αντιπροσωπιών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα κατά την άποψή μου είναι χαμηλός ο κίνδυνος αλληλεπικαλύψεων. Και όταν εντοπιστούν συγκεκριμένες δράσεις, πραγματικά μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι τότε δεν υπάρχει απόλυτος κανένας κίνδυνος αλληλεπικάλυψης. Πρόεδρος, ακούσατε οι τρεις εμπειρογνώμονες τι συζήτηση έγινε, τι είπαν οι βουλευτές της Επιτροπής μας. Θα σας δώσω λοιπόν στην καθεμία 1,5 λεπτό για να μπορέσει να πείτε στο δυνατόν περισσότερα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είπε ένα από του ομιλητέ ότι η μετανάστευση ε, αντιμετωπίζεται ω κάτι αρνητικό αυτή τη στιγμή. Αλλά για τους μετανάστες ε, ε, είναι πιστεύω κάτι πολύ θετικό. Δηλαδή για τη μείωση της φτώχειας είναι ίσως ο ταχύτερος τρόπος επίτευξε αυτού του στόχου. Γιατί λοιπόν αντιμετωπίζετε μετανάστευση ω κάτι αρνητικό. Οι μετανάστε φταίνε το ότι βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει, πιστεύω, με γενικότερες ε, προκλήσεις ε, προς την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Δηλαδή, πώς ρυθμίζουμε τις αγορές εργασίας της Ένωση, πώς μεταρρυθμίζουμε τα κοινωνικά ασφαλιστικά συστήματα, οι ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι αλληλέγγυες, ε, δείχνουν ανοχή, ανεκτικότητα. Μπορεί ο κόσμος να χρησιμοποιήσει τις ε, δυνατότητες που του παρέχουν τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αξιοποιήσει τα ταλέντα του. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η αρνητική αντίληψη, η οποία επεκτείνεται και πηγαίνει και στους αναπτυξιακούς στόχους. Όταν δηλαδή η ανάπτυξη θεωρείται ένας τρόπος για να αντιμετωπιστούν ε, οι βαθύτερες αιτίες της μετανάστευσης, αυτό μπορεί να είναι καλό σε κάποιε περιπτώσει, αλλά πιστεύω ότι είναι και σφάλμα να θεωρούμε ότι η ανάπτυξη σημαίνει ότι η μετανάστευση από τι τρίτε χώρε πρέπει να σταματήσει. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Μπορεί να, ε, να είναι διαφορετικοί άνθρωποι που θα μεταναστεύουν, γιατί είναι αρκετά δαπανηρή η όλη διαδικασία, αλλά συμβαίνει παρόλα αυτά. Και σε σχέση με αυτό που είπα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, ίσω αυτοί οι άνθρωποι επιλέξουν έναν άλλο προορισμό που, τους, ε, που θα του δεχθεί πιο εύκολα. Και η πολιτική κυρίως έχει να κάνει με την επισδοχή, την επιστροφή. Δεν ξέρω αν αυτό όμως είναι και η βέλτιστη αντιμετώπιση ή προσέγγιση. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ που μου ξαναδώσετε το λόγο. Θέλω να τονίσω λίγο περισσότερο. Αυτό το εργαλείο Πολιτική για την ανάπτυξη που μπορεί να βοηθήσει στη λήψη πιο δίκαιων και καλύτερων αποφάσεων. Δεν είναι όμω μόνο ένα εργαλείο, είναι και μια υποχρέωση. Μια υποχρέωση η οποία έχει να κάνει με τη γαμαδοδέλτα εσωτερικών υποθέσεων, για τι αποφάσει δηλαδή που πρέπει να λαμβάνονται στην εξωτερική διάσταση τη πολιτική μετανάστευση. Όταν λοιπόν μιλάμε για κριτήρια για τον καθορισμό του τι πρέπει να χρηματοδοτηθεί και από ποιο μέσο, όποια και αν είναι αυτά τα κριτήρια, η ανάπτυξη είναι ένα από αυτά τα κριτήρια το ότι θα πρέπει να είναι συνεκτικέ και συνεπεί με του αναπτυξιακού στόχου, αυτέ οι αποφάσει και θα πρέπει να βλάπτουν τη διαδικασία αυτή είναι μια υποχρέωση με βάση τη συνθήκη τη Λισαβόνα και αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και ήθελα να το τονίσω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, συνδέονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυτά που προείπα και επίση τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υποχρέωση και αδιαπραγμάτευτο ζήτημα. Εξού και δεν υπάρχει παράνομο ε, ανθρώπινο ε, αυτή η έννοια δεν υφίσταται. Το θέμα είναι να συσχετίσουμε αυτές τις δύο συνιστώσεις και να μην μείνει ε, μια στόχη, την ανθρώπινη δικαιότητα μόνο στο αναπτυξιακό πεδίο. Νομίζω ότι μπορούμε τι αναπτυξιακέ ανησυχίε και παραμέτρου να τι συμπεριλάβουμε σε όλε τι σε άλλου τομεί πολιτική. Είναι πολύ καλό που ε, έγινε αυτή η πρόταση για έναν εσωτερικό διάλογο και με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και άλλες επιτροπές ε, και σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Η τρίτη προσκεκλημένη είναι σας ευχαριστώ που μας ξαναδείτε το λόγο. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ πρόσδεκτες οι διευκρινήσεις που δόθηκαν σε σχέση με το τι χρηματοδοτείται στο πλαίσιο των εσωτερικών ε, ταμείων και τι ε, στο πλαίσιο της εξωτερικής διάστασης. Εμείς θα θέλαμε να το δούμε και εγγράφως αυτό και στα σχέδια δράσης, τα μελλοντικά. Επίσης είναι σημαντικό και την έκκληση προς την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς αυτό το έργο για την προστασία των ε, προσφύγων και για τη μετανάστευση στις τρίτες χώρες να είναι πιο ορατό. Η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη μόνο την διαχείριση της μετανάστευσης προς την Ευρώπη γνωρίζει. Το ότι όμως η Ένωση δαπανά πόρους σημαντικούς για συνεργασία με τρίτες χώρες και στηρίζει τους μετανάστες, βοηθά τους πρόσφυγες, προστατεύει τους πρόσφυγες, είναι κάτι που δεν είναι καθόλου γνωστό. Και νομίζω ότι για να αντιμετωπιστεί η ξενοφοβία και ο ρατσισμός είναι κάτι που πρέπει να προβληθεί. Είναι ένα σημαντικό καθήκον, πιστεύω, για την ε, Κομισιόν και για το Κοινοβούλιο. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ όλες σας για αυτή τη συζήτηση. Δεν ξέρω τι νιώθετε εσείς, αλλά εγώ πραγματικά νιώθω μεγάλη απογοήτευση που δεν μπορέσαμε να έχουμε περισσότερο χρόνο να ακούσουμε περισσότερα σχόλια στο πλαίσιο αυτή τη συζήτηση. Ίσως θα πρέπει να διοργανώσουμε μια ακρόαση για αυτό το θέμα. Ίσως θα πρέπει να θέσουμε αυτό το ζήτημα στους συντονιστές. Now we come to something very, very important. Περνάμε τώρα σε κάτι το πολύ σημαντικό. Ε, χρηματοδοτικά μέσα για την αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι η δεύτερη ανταλλαγή απόψεων που θα έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση συνεργασίας. Τον Φεβρουάριο είχαμε την πρώτη συζήτηση επί τη βάση της μελέτης της ECDPM για τα χρηματοδοτικά εξωτερικά μέσα από τότε. Η εσωτερική μας συζήτηση έχει προχωρήσει αρκετά. Η ομάδα εργασίας DCI συναντήθηκε δύο φορές και συζήθηκε συγκεκριμένα θέματα και προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συζητήσεις έγιναν και με άλλες επιτροπές που ασχολούνται με τέτοιου είδους θέματα. Ιδιαίτερα με την ΑΦΕΤ, η οποία είναι και η επί της ουσίας, θα έλεγα, επιτροπή. Έχουμε τη δυνατότητα τώρα να προχωρήσουμε σε ε, βάθος στη συζήτηση αυτή, να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα δώσω το λόγο πρώτα στον εισηγητή μας και μετά θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές. Εισηγητής μας αυτό το ε, ε, πολύ σημαντικό θέμα είναι ο Τις Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι πρόκειται για τη δεύτερη ανταλλαγή απόψεων. Δεν έχω την Ιρλανδική σαν γλώσσα εργασίας και θα μιλήσω στα αγγλικά. Είχαμε τη συζήτηση αυτή σε ένα δύσκολο οικονομικό πλαίσιο για την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο υπάρχουν σκληρές πολιτικές επιθέσεις στις ίδιες τις αρχές της αναπτυξιακής βοήθειας, αλλά ακόμα και η βοήθεια και η στήριξη του κοινού παρότι παραμένει ισχυρή μειώνεται. Και ε, το να μειώνει κανείς τον αναπτυξιακό προϋπολογισμό φυσικά ευνοεί τους αριθμούς του κρατικού προϋπολογισμού και εκεί έχουμε ένα θέμα. Ευτυχώς ε, έπεσε η κυβέρνηση στη χώρα μου, ευτυχώς λέγω χτες. Και έτσι η μείωση κατά ένα δις, κατά 750 εκατομμύρια μάλλον, ε, που προεβλέπεται να υπάρξει ε, απεκλείστη τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα, αν και δεν είμαι πολύ αισιόδοξο. Η κατάσταση λοιπόν δεν είναι πάρα πολύ εύκολη και θα πρέπει να δούμε αν ο προτινόμενος προϋπολογισμός για την ανάπτυξη για τον DCI τα 23,300 εκατομμύρια, 23 εκατομμύρια θα επιβιώσουν στο τέλος, ίσως να είναι και λίγο λιγότερα. Στον αναπτυξιακό κόσμο βέβαια η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη. Υπάρχει οικονομική ανάπτυξη στους περισσότερους ε, χώρους, στις περισσότερες περιοχές. Υπάρχουν θέματα δημοκρατίας βέβαια και εκδημοκρατισμού, αλλά όλα αυτά συμβαίνουν σε πλαίσια τεράστιας κοινωνικής ανισότητας και άλλα πολλά σοβαρά προβλήματα όπως οι συνέπειες των ε, κλιματολογικών αλλαγών. Έχουμε μία συζήτηση λοιπόν σε ένα πλαίσιο θα έλεγα πολιτικό διόλου εύκολο και αυτό μας ρίχνει τεράστιες ευθύνες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προσπαθήσει να αξιολογήσει καλύτερα την ισορροπία ανάμεσα στις αξίες που την εμπνέουν, στα συμφέροντά της και στις πολιτικές της θα πρέπει εμείς να συμπεριλάβουμε την βασική ιδέα, τη βασική αρχή της συνολικής ανάπτυξης, της ολοκληρωμένης ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και αυτή η ιδέα θα πρέπει να είναι χρήσιμη για όλους και ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι αντιμετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες ενσωμάτωσης στην ε, κοινωνία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στις βαθιές κοινωνικές απαραίτητες αλλαγές και φυσικά και στα θέματα διασφάλισης προμήθειας τροφίμων. Όλα αυτά μπορούμε να τα πετύχουμε τα επόμενα δέκα χρόνια, αλλά έχουμε τεράστιες δυσκολίες λόγω των κλιματιλογικών αλλαγών, της μείωσης των αρρωσίμων γεών στον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν ορισμένα θέματα λοιπόν τα οποία θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας σήμερα. Ζητώ συγγνώμη για τα αγγλικά μου προς τους διερμηνείς λέει ο μιλητής αλλά συνεχίζει στα αγγλικά. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα θέματα που πρέπει να δούμε και το ένα είναι η προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το μελλοντικό αυτό μέσο αναπτυξιακής συνεργασίας θα πρέπει να δείχνει με καλύτερο τρόπο το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματώνει τις δυνατότητες τις οποίες έχει σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ένας απλός δωρητής, Αυτό που έχει σημασία είναι να συνδυάσει την βοήθεια αυτή με το πολιτικό βάρος το οποίο έχουν οι 27 χώρες μέλη. Και το βάρος αυτό είναι υπέρημον για να αντιμετωπίσουμε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτους δικαίου, δημοκρατίας, βελτίωσης της κατάστασης στα λεγόμενα εύθραυστα κράτη, και θα έλεγα ότι εμείς θα πρέπει να είμαστε αυτοί που κηρύσουν ή μάλλον να υπερασπιστούμε αυτούς οι οποίοι υποφέρουν από κοινωνικές ε, συγκρούσεις και ανισότητες. Το θέμα λοιπόν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα πλαίσια της ανάπτυξης είναι κάτι το οποίο βοηθιέται από την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία μπορεί να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα δεν είναι να ασχολούμαστε μόνο με κάποια κλειστά θέματα, θα έλεγα θεματολογικά μάλλον περιορισμένους τομείς. Θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε σφαιρικά το πρόβλημα. Και θα πρέπει έτσι, αν το κάνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να επικοινωνήσει καλύτερα και αποτελεσματικότερα. Αυτό το έλεγε για πρώτη φορά και ο ΑΣΑ στο σχέδιό του ε, για τον τομέα που μας ενδιαφέρει ήδη από το 2007. Το ίδιο πρέπει να πούμε και τώρα. καλύτερος και περισσότερος συντονισμός. Τώρα, υπάρχει λόγος να στρέψουμε τη βοήθειά μας την αναπτυξιακή σε αυτούς οι οποίοι έχουν περισσότερες ανάγκες. Χώρες δηλαδή οι οποίες είναι πτωχές χαμηλών εισοδημάτων ή μεσαίων χαμηλών εισοδημάτων και η πρόταση η οποία περιλαμβάνεται εδώ στο σχέδιο για το DCI είναι μια καλή θα έλεγα πρόταση και προϋποθέτει σωστούς ρυθμούς ανάπτυξης. δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά ένα κριτήριο όπως το ΑΕΠ, ενώ θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τον δείκτη της ανθρώπινης ολοκλήρωσης ή ανάπτυξης να δούμε τα θέματα της ανάπτυξης με πιο θετικό και προσδιορισμένο τρόπο. Secondly, differentiation, a clear cut from 100 to 0, I would say, let it be a phased approach. Θα πρέπει να μην υπάρχουν απότομες αλλαγές, να υπάρχει μια σταδιακή κλιμάκωση προβλέψιμη που να συνοδεύεται από ισχυρό πολιτικό διάλογο με τις αρμόδιες περιφερειακές και εθνικές αρχές των χωρών που δεν θα μπορούν να είναι πλέον επιλέξιμες. Και αναφέρομαι σε χώρες όπως Ινδία, Κίνα, Βραζιλία ε, και ενώ θα σταματήσουν τέτοιου είδους γεωγραφικές ε, ε, προσπάθειες βοήθειας θα συνεχιστούν σε επίπεδο συγκεκριμένων τομέων παρέμβασης βέβαια Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φιλόδοξους στόχους για τις συνέπειες των κλιματολογικών αλλαγών. Είναι λογικό να συμπεριλάβουμε τους τομείς αυτούς στην αναπτυξιακή μας πολιτική. Η πρόταση όμως για το DCI περιλαμβάνει προτάσεις επιλέξιμες και προγράμματα υποστηρίξιμα, αλλά ε, όλα αυτά φυσικά πρέπει να έχουν άμεση συσχέτιση και με τις κλιματολογικές αλλαγές και το περιβάλλον. Θα πρέπει λοιπόν η χρηματοδότηση για μέτρα τα οποία συνδέονται αυστηρά όμως με τις κλιματολογικές αλλαγές να είναι επιπλέον, να είναι συμπληρωματική. Θα πρέπει να υπάρξει η αρχή της προσθετικότητας έτσι ώστε να συμπεριληφθεί η κλιματολογική ε, θα έλεγα διάσταση στο DCI. Θα πρέπει επίσης να υπάρξουν επαρκείς οικονομικές παρεμβάσεις στον τομέα των βασικών κοινωνικών αναγκών. Εμείς είχαμε βάλει το όριο του 20% και γίνεται δεκτό. Αλλά είναι κάτι το οποίο εξηγείται, τεκμηριώνεται ήδη από την συνάντηση την κοινωνική κορυφής του 1995. Είναι φυσικά απαραίτητο για να πετύχουμε τους περαιτέρω στόχους μας να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες. Και στην πρόταση για τον DCI και στην πρόταση για τις αλλαγές στην ατζέντα η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει την έννοια της κοινωνικής συμπερίληψης ε, και της ε, προσωπικής ολοκλήρωσης και ανάπτυξης. Κατανοώ τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σαν πολιτικός και εγώ είμαι υπέρ της ε, ευελιξίας, αλλά θα πρέπει όμως να μην χάνουμε εδώ την δυνατότητα ελέγχου. και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν καλύτερα κάποιοι δείκτες, ε, σαν παράδειγμα αντί να μιλήσουμε γενικά για κοινωνική συμπερίληψη, να χρησιμοποιήσουμε στατιστικά επαληθεύσιμα στοιχεία κοινωνικής κάλυψης. Αν οι αναπτυξιακές πολιτικές θέλουμε να είναι ωφέλιμες, τότε θα πρέπει να επιδοτήσουμε τις προσπάθειες μέσω δανείων, μέσω επιδοτήσεων που οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη έτσι ώστε να μπορέσει ε, η κατηγορία αυτή του πληθυσμού να ενταχθεί στην οικονομία. Οι προτάσεις που ακούστηκαν μέχρι τώρα είναι καλές. Έβδομο σημείο. Στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση με την βοήθεια την έκτακτη, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη. Βασιζόμαστε στη διατύπωση του ισχύοντος DCI. Όμως, θα πρέπει να συνδέσουμε καλύτερα την βοήθεια, την έκτακτη, την σωστική θα έλεγε κανείς, με την αναπτυξιακή βοήθεια, σε συνεργασία με, τους, με τις τοπικές σε συνεργασία με τις ΜΚΟ της αναπτυξιακές, θα πρέπει να βρούμε μέτρα τα οποία να είναι συμβατά μεταξύ τους και να καλύπτουν γρήγορα τις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν. Και υπάρχουν και κάποια άλλα προγράμματα όπως το Παναφρικανικό πρόγραμμα ενός δις που προβλέπει το DCI. Καλό είναι να δοθεί ένα δις για να μπορέσει κανείς ε, να χρηματοδοτήσει τμήματα της ευρωαφρικανικής στρατηγικής ή της αφροευρωπαϊκής καλύτερα να το πω στρατηγικής. Βέβαια οι στόχοι αυτοί είναι ο λίγον δυσδιάκριτοι και απαιτείται μεγαλύτερη ευκρίνεια για το τι είναι το Παναφρικανικό πρόγραμμα. Τώρα για το Κοινοβούλιο. Υπάρχει συζήτηση και σε επίπεδο της κοινωνίας των πολιτών για τα επι, επιμέρους θεματολογικά προγράμματα. Σαν βουλευτής εγώ ε, θα πρέπει να ζητήσω να αναγνωριστεί με καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο ο ρόλος του Κοινοβουλίου, έτσι ώστε τα κοινοβούλια να μπορούν να έχουν οι υπόλογες τις κυβερνήσεις τους που εφαρμόζουν αυτού του είδους τα μέτρα. Και τέλος, συνοχή. Μιλήσαμε για τη συνοχή σε σχέση με τους αναπτυξιακούς στόχους Νομίζω ότι εδώ ε, η παρουσίαση που γίνεται είναι λίγο αντίστροφη αυτής που χρειαζόμαστε. Οι αναπτυξιακές πολιτικές θα πρέπει να είναι λέει συμβατές με τις υπόλοιπες πολιτικές. Δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα. Όλες οι πολιτικές θα πρέπει να είναι συμβατές με την μείωση της ένδυας στον κόσμο. Τέλος θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όλους να μην κάνουν και πάρα πολλές τροπολογίες σε λεπτομέρειες και να μην καταστήσετε την έκθεσή μου χριστουγεννιάτικο δέντρο. Thank you, Ευχαριστώ για την εξαιρετική εργασία την οποία κάνετε και για το γεγονός ότι Τώρα τονίζεται περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα που πρέπει να οθήσουν την ανάπτυξη ε, είναι οι πρωτοβουλίες της ήπιας επίδειξης δυνάμεως και τώρα ο Γκάι Μίτσελ που είναι ο εισηγητής για το ΕΛΚ και ο προηγούμενος ε, εισηγητής ε, για το DCI. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω λίγα λόγια σχετικά με το θέμα και θα συμβιβαστώ μιλώντας αγγλικά. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω για τη δουλειά που έγινε. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι το Κοινοβούλιο σωστά προσήγησε το θέμα αυτό και πρέπει να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, δηλαδή να μην προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο και έναν Άγιο Βασίλη, αλλά το Κοινοβούλιο πρέπει να εξασφαλίσει ότι θα ακουστεί η φωνή του Κοινοβουλίου, διότι οι ψηφοφόροι προσπαθούν να μας διαχωρίσουν και χρειάζεται ε, κάποια κάποιο κίνητρο για να βρούμε περισσότερα κοινά σημεία, κοινώς αποδεκτά σημεία. Όσον αφορά το DCI πιστεύω ότι θα πρέπει να καταρτιστούν στόχοι διαφάνειας και να είναι υπόλογος ο οργανισμός διότι χωρίς αυτές τις ε, λεπτομέρειες δεν θα προχωρήσουμε. Αναρωτιέμαι όμως ότι, τι έγινε στο παρελθόν, επιτύχαμε το στόχο του 20%, τι καταφέραμε, διότι ξέρω ότι αυτό είναι βασικό θέμα και θα πρέπει να ανανεώσουμε ε, την, ε, τους αναπτυξιακούς στόχους και ε, πρέπει να πούμε ότι είμαστε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στα κράτη-μέλη αλλά ε, βλέπουμε ότι και αν μειώνεται η συνδρομή μας στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων δεν θα πρέπει να μειωθούν πέραν ενός συγκεκριμένου επίπεδου και γι' αυτό θα πρέπει να πούμε στα κράτη-μέλη ε, τι γίνεται θετικά στις υποανάπτυξη χώρες και να μην μιλήσουμε μόνο για απελπισία και χάος. Πρέπει να δούμε και τι θετικό επιτυγχάνεται και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω ότι θα πρέπει να προβληθεί. Ε, ο Bill Gates μίλησε για επιτυχίες, ε, οπότε πρέπει να ρωτήσουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ποιες είναι οι επιτυχίες μας, τι έχουμε επιτύχει και πιστεύω ότι ένα από τα θέματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε πέραν αυτών που είπε ο Τάις ε, για την Αφρική ε, είπα, μίλησε για μια χρηματοδότηση ενός δισεκατομμύριου αλλά πρέπει να ξέρουμε πώς θα χρησιμοποιηθεί και πρέπει να υπάρχει σωστή αντιμετώπιση. Δηλαδή υπάρχει οικονομική ασφάλεια την ε, οποία επιτυγχάνουν οι οικογένειες στον ανεπτυγμένο χώρο ε, με ε, μεγάλες οικογένειες και ιδίως με αγόρια. Ε, εάν υπάρχουν περιοχές όπου εάν διαπιστωθεί ότι το παιδί δεν είναι αγόρι τότε διακόπτεται η εγκυμοσύνη και εάν φτάσει στο, στην ολοκλήρωσή της υπάρχει γενοκτονία των ε, θηλυκών νεογνών ε, και πιστεύω ότι όλα αυτά είναι ένα οικονομικό βάρος διότι στην περίπτωση μεγάλες οικογενειών οι μεγάλες οικογένειες πιστεύουν ότι όσα περισσότερα παιδιά έχουμε τόσα περισσότερα παιδιά θα μας φροντίζουν στα γεράματά μας. Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή να σας παρουσιάσω ένα σύντομο έγγραφο επ' αυτού, ε, διότι και εμείς έχουμε αντιμετωπίσει τις ίδιες καταστάσεις στο παρελθόν. Και μην νομίζουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα διαφορετικό κόσμο. Υπάρχουν ε, μικρές επιχειρήσεις ε, που πολλούν οποροκυπευτικά, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα ή ε, πουλούν ε, ρουχισμό. Εάν ε, λοιπόν χρειαστεί να να δανειστούν για να ξεκινήσουν μία επιχείρηση ε, πάνε σε ένα χειροδανιστήριο, καταστρέφονται οικονομικά για να αποπληρώσουν ε, και γι' αυτό στις υποανάπτυξη χώρες ε, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα προωθήσεως των γυναικών και γι' αυτό καταφεύγουν στις μεγάλες οικογένειες. Δεν σας μιλώ εδώ εκ του προχείρου. Έχω έχω ε, ε, έχω εξετάσει την περίπτωση αυτή. Ε, μιλάμε για ασφάλεια 10-20% δολάρια για άτομα που ζουν με 99 cent είναι τεράστια ποσά και ίσως θα πρέπει να επιζητήσουμε να διελευκάνουμε άλλα θέματα, δηλαδή να εξετάσουμε πόσο θα ενθαρρύνουμε μία κυβέρνηση, πολλές κυβερνήσεις για ένα πιλωτικό πρόγραμμα να δούμε αν μπορούμε να στηρίξουμε τις ασφάλειες κατά τρόπον ώστε όσοι μπορούν να δημιουργήσουν μία μικρή επιχείρηση που θα τους βοηθήσει να επιβιώσουν μπορούν να, να ασφαλιστούν και να δώσουν ένα μέρος του κεφαλαίου κεφαλαίου για την ασφάλιση αν κάποιος άλλος τους ε, ε, επιδοτήσει για ένα άλλο μέρος του κεφαλαίου τους. Βέβαια δεν πρέπει να τα κάνουμε στο ποδάρι, πρέπει να τα εξετάσουμε και να δούμε αν ε, υπάρχει δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει εάν αυτοί οι οποίοι δεν εξαρτώνται από μεγάλους αριθμούς και από μεγάλα κεφάλαια μπορούν επίσης να βοηθηθούν. Να δούμε δηλαδή νέες ιδέες, νέα θέματα και ε, αυτό θα είναι κάτι που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Επίσης ο Τάις αναφέρθηκε στη συνεκτικότητα και συζητήσαμε τη συνεκτικότητα στη συνάντηση με τους συζητητές την περασμένη, την προπερασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι ε, ε, είδαμε ότι διάφοροι συνάδελφοι ε, μπόρεσαν να συντονιστούν, να επισημάνουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να παρακολουθεί καλύτερα την τεράστια χρηματοδότηση του, των 5 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Θα μπορούσαμε μάλιστα να την αυξήσουμε ε, τη χρηματοδότηση αυτή σε 30 δισεκατομμύρια. Σκεφτείτε τι θα μπορούσαμε να επιτύχουμε με τα ποσά αυτά. Άρα κατά κάποιον τρόπο πρέπει να συνεργαστούμε με τα εθνικά κοινοβούλια διότι δεν επηρεάζουμε τις κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το γνωρίζει. Εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεργαστούμε με τα Εθνικά Κοινοβούλια για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει αυτή η πρόοδος και δεν ξέρω πώς αυτό θα επιτευχθεί αλλά όπως είπε ο Τσάρλς θα πρέπει να υπάρχει κάποια συνεργασία επί του θέματος πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το DCI πράγμα το οποίο θα γίνει μόνο αν γίνει ένας απολογισμός των ε, παρεμφερών προηγουμένων δράσεων ε, να ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος ε, και τι έχει γίνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, πολύ ενδιαφέρουσες και νέες ιδέες. Ο Σάλς Γκέρενς είναι ο επόμενος ε, ομιλητής, ο συγκητής από τη δική του ομάδα και εγώ θα εκπροσωπήσω εν συνεχεία τη δική μου ομάδα. Γιατί και εγώ έχω να πω κάποια πράγματα, ο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος διότι δεν άκουσα την παρουσίαση του ΤΕΙΣ, επειδή έπρεπε να συμμετάσχω σε μια άλλη συνεδρία που γίνεται παράλληλα και αφορά την Συμφωνία Άκτα. Θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με αυτά που είπε ο Γκέι Μίτσελ. Νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον μας να δούμε πώς επηρεάζει η πολιτική τη Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά την πολιτική αναπτυξιακής βοήθειας. Όταν επικεντρωνόμαστε στο DCI, ε, πιστεύω ότι είμαστε λίγο κοντόθωροι ναι, σημαντικό είναι ε, ως ε, μέσο. Πρόκειται για τις εκατομμύρια που θα δαπανηθούν. Αλλά πρέπει να δούμε και την συνεκτικότητα των πολιτικών και των δράσεων της ε, Κομισιόν και των κρατών μελών. Εμείς ως ε, Κοινοβούλιο θα πρέπει αυτό το διπλό ρόλο και της παρακολούθησης και της πολιτικής όθησης να φροντίσουμε να τον διενεργούν και τα Εθνικά Κοινοβούλια αλλά και εμείς. Στην τελευταία συνεδρίαση των συντονιστών ε, και ο Γκέι και εγώ προτείναμε τη σύνταξη μιας έκθεσης πρωτοβουλίας για αυτό το όλο ζήτημα. Όπου ένα μέλος της Επιτροπής μας και ένα μέλος κάποιου Εθνικού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να κάνουν ένα απολογισμό της κατάστασης και να διατυπώσουν προτάσεις, υποδείξεις για την πολιτική της αναπτυξιακής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι είναι ο συνθετικός κρίκος που λείπει από την αλυσίδα. Αν δεν υπάρχει κοινοβουλευτικό έλεγχος, κατά την άποψή μας δεν ε, κάνουμε επαρκές προσπάθειες να συντομινήσουμε καλύτερα τις διάφορες πολιτικές. Πάντοτε βέβαια παγρυπνούμε θέλουμε ε, τα κοινοβούλια των χωρών, των δικαιούχων να εφαρμόζουν πράγματα τα οποία θα πρέπει και εμείς να εφαρμόζουμε. Έχω πει στον ΤΕΙΣ, αλλά θέλω να το ξέρετε κι εσείς, ότι είμαι αρμόδιος για την μελλοντική ατζέντα για την ανάπτυξη, το θεματολόγιο για την ανάπτυξη. Θα προσπαθήσω με τον ΤΕΙΣ να μην ε, ε, επαναλαμβάνει ο ένας τις του άλλου. Θα διερευνήσω δηλαδή κάποιες διόδους και κάποιες άκουσε τις οποίες δεν έχει, με τις οποίες δεν έχει ασχοληθεί στην έκθεσή του ο για να συμπληρώνει η μία έκθεση στην άλλη και όχι να επικαλύπτονται. Κατά τα λοιπά είναι πολύ σημαντικό το έργο του ΤΕΙΣ για την Επιτροπή μας και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Ε, thanks, Σε ευχαριστώ, Σάρλ. Εγώ λοιπόν τώρα ο σκιώδης εισηγητής για την ομάδα ECR και όχι ως πρόεδρος σας, πρόεδρός σας, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Τέις για την πολύ καλή του δουλειά και αυτή που έχει ήδη κάνει και αυτή που θα κάνει στο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους οι οποίοι προτείνουν νέε ιδέε για το πώ πρέπει να προχωρήσουμε. Αλλά νομίζω ότι καλό θα ήταν να κάνουμε μια μικρή στάση και να διερωτηθούμε γιατί βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση και προσπαθούμε να ε, προβάλλουμε νέε ιδέε. Όχι γιατί απέτυχαν όλε οι ιδέε μα μέχρι τώρα, αλλά γιατί όλε οι πρωτοβουλίε επέτυχαν. Ο Σάρλ ε, ασχολείται με όλο αυτό το ζήτημα ε, της, του θεματολογίου για την αλλαγή, Agenda for Change, και ένα από τα στήματα που τίθενται είναι τι θα κάνουμε με τις χώρες μεσαίου εισοδήματο. Τι θα κάνουμε, θα διακόψουμε τις διμερείς μας σχέσεις με αυτές τις χώρες και θα τις αφήσουμε να σαπίσουν ε, οι φτωχοί σε αυτές τις χώρες ή θα υποχρεώσουμε αυτές τις χώρες να φροντίσουν για τους φτωχούς τους. Θα το συζητήσουμε και αργότερα, μία τουλάχιστον, στη νομογραμματότηση για τη Λατινική Αμερική. Διερωτώ με και χρησιμοποιώ και τη φαντασία μου αυτή τη στιγμή. Διερωτώ με λοιπόν μήπως θα μπορούσαμε να βάλουμε κάποιες προποθέσεις και κάποιους όρους, ώστε όταν έχουμε να κάνουμε με χώρες ε, μέσω εισοδήματος, ε, με υψηλή όμως κατά κεφάλιν ανάπτυξη, Να υπάρχουν λοιπόν κάποιοι όροι, κάποιες προϋποθέσεις, είτε μέσω των εμπορικών μας σχέσεων με αυτές τις χώρες, δηλαδή ή θα φροντίσουν τους φτωχούς τους με έναν τρόπο που εμείς κρίνουμε αποδεκτό, ή θα υιοθετήσουμε ένα λιγότερο ευνοϊκό εμπορικό καθεστώς με αυτές τις χώρες. Ή στο πλαίσιο του DCI να δούμε μήπως μπορούμε και εκεί να εντάξουμε αυτό το στόχο. Και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που έχει τρεις φορές το μέγεθος της Παγκόσμιας Τράπεζας στο κάτω-κάτω. Εμπορική τράπεζα είναι. Δεν χρηματοδοτείται από το φορολογούμενο. Μήπως λοιπόν και μέσω αυτής της τράπεζας, όπως χρησιμοποιούμε την Παγκόσμια Τράπεζα, θα μπορούσαμε να βάζουμε προϋποθέσεις για ε, την δανειοδότηση αυτών των χωρών. Δηλαδή να μπαίνει όρος ότι θα θετήσουν ε, ε, προγράμματα για να βοηθήσουν ε, τους φτωχούς, αυτούς που ζουν στις παραγκουπόλεις, παραδείγματος χάρη. Αλλιώ τι θα κάνουμε, θα αφήσουμε αυτές τις χώρες ε, όπω έχουν, οι φτωχοί να φτωχαίνουν περισσότερο και οι πλούσιοι να πλουτίζουν περισσότερο. Ένα αυτό. Δεύτερον, δικαιώματα ιδιοκτησίας. Πώς το DCI δηλαδή θα εντάξουμε μία μέθοδο που θα μας επιτρέψει να χρησιμοποιούμε τη δημιουργία υποδομών, το capacity building, για να βοηθούμε την καταχώρηση ε, των ε, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, ε, των επιχειρήσεων, πώς μπορούν να δημιουργήσουν ένα μικρό συνταξιοδοτικό πρόγραμμα, πώς μπορούν να λειτουργούν μια μικρή επιχείρηση την οποία έχουν συστήσει και ούτω καθεξής. Είμαστε σε μια διαδικασία αλλαγή και πρέπει να τα διερευνήσουμε όλα αυτά. Και λέω ότι έχουν υπάρξει επιτυχή παραδείγματα. Υπήρξαν ανεψόμενε χώρε που κατάφεραν, που πλουτίζουν και που ε, αναδύονται και αναπτύσσονται. Και εμεί ω μεγαλύτερο ε, χρηματοδότη, δωρητή, ε, έχουμε συνεισφέρει σε αυτό και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι θα πρέπει να είμαστε αυτάρες. Και έχουμε ε, τον Bill Gates, έναν από τους πλησιότερους ανθρώπους στον κόσμο, που θα τον αφήσουμε να μας λέει ε, πόσο ωραία τα έχουμε καταφέρει για την ε, παραγωγή και την διανομή προγραμμάτων. Ο Bill Gates μας είπε, εμάς, ότι χάρη στη δουλειά που έχουμε κάνει σήμερα ζουν 6 εκατομμύρια παιδιά που αλλιώς θα είχαν πεθάνει ή ασθενεί με ε, λονοσία και εγώ δεν ξέρω πόσοι θα είχαν πεθάνει. Γιατί δεν μα τα λέει αυτά η Κομισιόν και περιμένουμε να τα πει ο Bill Gates. Γιατί η Κομισιόν δεν έχει στοιχεία να μα πει πόσο καλά τα πήγε ή τα πήγαμε εμεί για να μπορούμε να ενημερώσουμε το φορολογούμενο. Να τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ορίστε, οι επιτυχίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα στοιχεία. Πόσοι άνθρωποι σήμερα που θα είχαν πεθάνει, αν δεν είχαμε κάνει ό,τι κάναμε, ζουν σήμερα. Πόσα παιδιά σήμερα βρίσκονται στο σχολείο ή ε, φοιτούν, δεν θα είχαν εκπαίδευση αν δεν είχαμε κάνει αυτά που κάνουμε, πόσα άτομα μπορούν να συλληφθούν στο νοσοκομείο, που υπάρχει εκτρισμό κτλ. κτλ. Δεν θα έπρεπε να τα λέμε εμεί αυτά. Μα τι συμβαίνει. Ποιο είναι το πρόβλημα με την Κομισιόν που δεν μα λέει τα στοιχεία και πρέπει να βασιζόμαστε σε έναν Αμερικανό εκατομμυρίουχο που θα μα πει τι κάνουμε εμεί. Πραγματικά έχω συγχυστεί πάρα πολύ με αυτό. Και γι' αυτό ειλικρινά ζητώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εκπονήσει ένα έγγραφο στο οποίο θα απαριθμεί τις επιτυχίες μας για να το ε, παρουσιάζουμε στους φορολογουμένους μας. Τουλάχιστον εγώ στη δική μου εκλογική περιφέρεια που με ρωτάνε γιατί δαπανάτε τα χρήματά μας, προς ποιους στόχους. Χρειάζεται απάντηση. Αυτό είχα να πω. Ευχαριστώ. Ricardo, Ο Ρικάρντο τώρα θα λάβει το λόγο. On behalf <laughs> not here. Εκ μέρου ε, κανενό τέλο πάντων, λέει ο πρόεδρο. Ευχαριστώ πολύ κύριε πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Τέσ για τη δουλειά του. Πάρα πολύ σημαντική η έκθεση αυτή για την Επιτροπή μας. Άρα, αναμφίβολα επιτελεί τεράστιο έργο και είμαι βέβαιο ότι θα είναι θετικά τα αποτελέσματα. Ήθελα να πω στον πρόεδρο ότι δεν χρειάζεται να έρχεται ο Bill Gates για να μα ε, μιλήσει για την πολιτική ανάπτυξη. Είτε έρθει είτε δεν έρθει ο Bill Gates, ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Ευρωπαίοι πολίτε πώ έχει ε, λειτουργήσει η αναπτυξιακή πολιτική όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρουν οι πολίτε τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τη συνεργασία και την ανάπτυξη μια δέσμευση η οποία θα συνεχιστεί. Και υπάρχει έργο που έχει επιτελεστεί και θεωρώ ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες στην πλειονότητά του το γνωρίζουν αυτό το έργο και θα συνεχίσουν να το στηρίζουν και στο μέλλον. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια και μια ερώτηση. Από πού να αρχίσω. Ας ξεκινήσω με το ερώτημα. Η κατάσταση ε, των διαπραγματεύσεων για την πρόταση του νέου μέσου εταιρικής σχέσης Πώς έχουν τα πράγματα. Τι μπορείτε να μας πείτε, κύριε Σιγητά, πάνω σε αυτό. Και δύο-τρία σχόλια, δύο-τρεις σκέψεις ε, που έχουν να κάνουν ακριβώς με αυτές τις χώρες ε, μεσαίου εισοδήματος. Υπήρξε ε, διάσκεψη κορυφής στο Μπουσάν και εκεί μιλήσαμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Για παραγωγικότητα της βοήθειας, δηλαδή τι αποτελέσματα δίνει όπως εγώ τουλάχιστον ε, καταλαβαίνω τα πράγματα, δεν μπορεί να διακοπεί έφνης η βοήθεια προς κάποιες χώρες. Μπορεί να είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα που γίνονται στη χώρα από ένα μακροοικονομικό στοιχείο, από ένα νούμερο. Μη συγχαίουμε την πραγματικότητα με ένα μακροοικονομικό στοιχείο δηλαδή. Πιστεύω λοιπόν ότι με όλε τι χώρε από οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου, πρέπει να γίνει προσπάθεια. Μιλάω για όλε τι χώρε που αναλαμβάνω όλων των ε, περιοχών. Α κάνουμε phasing out, σταδιακή εξάλληψη, όχι απότομα να διακόψουμε τη βοήθεια που παρέχουμε σε κάποιε χώρε με μία αιτιολόγηση, λεγοντα ότι έχετε μία ανάπτυξη, έχετε αυτό το στοιχείο, αλλά όταν η πραγματικότητα στη χώρα και η δέσμευση που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση για αναπτυξιακή συνεργασία με τη χώρα αυτή, πρέπει να συνεχιστεί. Νομίζω ότι θα έπρεπε να επιλέξουμε μια πιο μετριοπαθή και βαθμιαία μετάβαση ε, που να ακολουθεί την κοινή λογική. Δεν είναι η συνεργασία, είναι κοινό νους. Πρέπει να υπάρξει μια ε, βαθμιαία έξοδος. Και σε ό,τι αφορά την προστιθέμενη αξία. Νομίζω ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία. Δηλαδή θέλουμε η βοήθεια να φτάσει σε αυτούς που τη χρειάζονται περισσότερο. Και επειδή αυτή είναι η δομή μέχρι τώρα που είχαμε και ε, λειτουργήσε θετικά μέχρι τώρα θεωρώ. Τα γεωγραφικά προγράμματα έχουν κάποιες ειδικέ οροφές. Παραδείγματο χάρη, όταν κλείσουν κάποια προγράμματα ε, σε κάποιες χώρες με μέσο εισόδημα, μήπως θα μπορούσαμε τους πόρους αυτούς να τους χρησιμοποιήσουμε και πάλι στις ίδιες χώρες ή σε άλλε χώρε τη ίδια περιοχή, ευρύτερη, που αντιμετωπίζουν τι ίδιε δυσκολίε. Δηλαδή, να γίνει ένα επαναπροσανατολισμό. Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνω, ξαφνική διακοπή βοήθεια με κάποιε χώρε δεν έχει κανένα, κατά την άποψή μου, αντίκρισμα. Και δεύτερον, ενίσχυση τη συνεργασία. Γιατί έχουμε πετύχει θετικά αποτελέσματα και μπορούμε να συνεχίσουμε να έχουμε αποτελέσματα εάν διατηρήσουμε αυτή τη δέσμευση. Δηλαδή, να παρέχουμε βοήθεια στις χώρες που το χρειάζονται περισσότερο και ε, επαναλαμβάνω να τους ε, παρέχουμε λύσεις και να αποχωρούμε βαθμιαία, όχι απότομα. Μήπως κάποιος άλλος συνάδελφος θα ήθελε το λόγο πριν δώσω τον λόγο στην Επιτροπή. Ο εκπρόσωπος λοιπόν της Επιτροπής. Ε, ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Μπέρμαν θύμισε το ευαίσθητο οικονομικό και πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο παρουσιάζουμε τις προτάσεις μας. Το πολιτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο των κρατών μελών θα παίξει ρόλο στις ε, διαπραγματεύσεις και θα ήθελα να χαιρετήσω το θάρρος και τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί στο τμήμα 4 ε, προβλέπουμε αυξήσεις και πιστεύουμε ότι το τμήμα 4 και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης νηστά προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πετύχουν έτσι καλύτερα τα προγράμματα που καθόρισε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και εφαρμόζει η Επιτροπή. Εγώ ο ίδιος είμαι πεπισμένος για την επιτυχία αυτού του σχεδίου. Είχα διατυπώσει πριν δύο χρόνια ε, ένα μικρό έγγραφο για την αναθεώρηση των στόχων της χιλιετίας στη Νέα Υόρκη. Είναι αλήθεια βέβαια ότι στο παρελθόν δεν μας άκουγαν τόσο πολύ και ζητούσαν να είμαστε πιο μετριοπαθείς. Θυμάμαι ότι η Κλέα Σόρτ πριν λίγα χρόνια έλεγε ότι ήμασταν οι χειρότεροι δανειστές στον κόσμο. Από τότε όμως άλλαξαν πολλά, ο χρόνος πέρασε και βελτιωθήκαμε χάρη και στη δική σας στήριξη και σήμερα είμαστε πολύ περήφανοι για τα προγράμματα τα οποία προσπαθούμε να προωθήσουμε. Υπόθηκαν μέχρι τώρα πολλά, θα ήθελα λίγα θέματα να θέσω. Πρώτον, τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την ανάπτυξη και τη σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εδώ υπάρχει σύγκληση, ε, θα έλεγα, και με το Συμβούλιο, όχι μόνο με το Κοινοβούλιο. Στον στόχο 1 βάζουμε ένα συγκεκριμένο, μια συγκεκριμένη αναφορά για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Έχουμε στο άρθρο 3 τις γενικές αρχές και στο πρώτο σημείο λέμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου αποτελούν το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο θα εφαρμοστεί η συμφωνία και το άρθρο 16 για την διακοπή της συμφωνίας λέγει ότι η βοήθεια μπορεί να διακοπεί στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει σεβασμός των ανωτέρων αρχών. Σχετικά τώρα με την συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της συνεργασίας αυτής. Βάλαμε στον κανονισμό μας την ανάγκη μιας μικτής ε, επικοινωνίας μάλλον θα έλεγα με, την, με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Πήραμε τα πρώτα μέτρα έτσι ώστε να γίνει πραγματικότητα. Βέβαια για να χορέψει κανείς χρειάζονται δύο χορευτές και γι' αυτό ζητάμε λοιπόν και τα κράτη-μέλη να κάνουν τις απαιτούμενες προσπάθειες για να μπορέσουμε να καταστήσουμε λειτουργική αυτή την πρόβλεψη και τον κοινό προγραμματισμό. Διότι εφόσον προγραμματίσουμε από πριν, τότε θα μπορέσουμε να υποφεληθούμε από τα ωφέλη σε εισαγωγικά της σωστής εφαρμογής της βοήθειας προς τρίτες χώρες. Τώρα, για την διαφοροποιούμενη αντιμετώπιση. Νομίζω ότι σταθήκαμε θαραλέοι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θελήσαμε να διαρρήξουμε τις σχέσεις μας με το παρελθόν. Πιστεύουμε ότι ορισμένες τρίτες χώρες είχαν πετύχει αρκετά πράγματα κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών και ότι θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας τις αναπτυξιακές αυτές εμπειρίες. Ε, προτείναμε λοιπόν τη σταδιακή αντιμετώπιση ορισμένων χωρών που δεν είναι πλέον επιλέξιμες σε διμερές επίπεδο, αν και θα συνεχίσουμε να διατηρούμε έναν πολιτικό, εμπορικό και θεματολογικό επιμέρους διάλογο με τις χώρες αυτές. Επειδή οι χώρες αυτές παραμένουν επιλέξιμες στο θεματολογικό πρόγραμμα ή στα περιφερειακά προγράμματα. Για αυτήν λοιπόν τη σταδιακή αντιμετώπιση αυτών των χωρών επιλέξαμε ένα συγκεκριμένο δίκτυο ο οποίο αναγνωρίζεται από όλους που είναι ο κατάλογος ε, για τη βοήθεια για την ανάπτυξη που ε, θα έλεγα ταξινομεί τις χώρες αυτές λέγοντας πως το σύνολο των χωρών ε, με μέσα εισοδήματα ή ανώτερα εισοδήματα θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σταδιακά σε φάσεις γιατί οι χώρες αυτές έχουν κάποιες δυνατότητες οικονομικές για να εφαρμόσουν κοινωνικές πολιτικές καταπολέμησης της ένδυας. Μιας και πρόκειται για μια μετάβαση, μια μεταβατική περίοδο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από εσωτερικές μελέτες δεν έκανε συγκεκριμένες προτάσεις λέγοντας ότι ναι ε, χρειάζεται διάλογος με τις χώρες αυτές αλλά μιας και πρόκειται για περιπτώσεις μεταβατικές, είπαμε ότι τα προγράμματα τα οποία λειτουργούν μέχρι το 2013 μπορεί να αναπτυχθούν μέχρι και το 2017 στις χώρες αυτές. Και τελικά οι χώρες αυτές οι οποίες ταξινομούνται με τον νέο τρόπο δεν εξαρτώνται από τη βοήθειά μας και οι επιπτώσεις της βοήθειάς μας ήταν ιδιαίτερως περιορισμένες σχετικά με τους εθνικούς τους προϋπολογισμούς. Είμαστε φυσικά σε, στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για επιμέρους πληροφορίες για το θέμα αυτό. Για τα θέματα της κοινωνικής προστασίας, είτε για την κοινωνική πρόνοια, είτε για την ασφάλεια υγείας, αυτά είναι προτεραιότητα για μας και θα είναι ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Θα κάνουμε μια ανακοίνωση πριν το τέλος του χρόνου και θα έχουμε την δυνατότητα να επανέλθουμε σε όλα αυτά. for that. Ναι, θα επανέλθουμε ε, διότι νομίζω ότι είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που έχεις να μας πεις και ε, θα θέλαμε να καταρτήσετε ένα σύντομο έγγραφο όπου θα λέτε ουσιαστικά ε, πόσους, ε, ε, πόσα άτομα τρέφουμε αυτή τη στιγμή, πόσοι εμβολιάζονται, πόσοι θεραπεύονται βάσει των δράσεών μας. Νομίζω ότι θα είναι πολύ επικοδομητικό για την έρευνά μας. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Charles Γκέρενς να παρέμβει τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω μία ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το πρόγραμμα Έρασμους διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να γδίσει τον έναν για να ντύσει τον άλλον. Δηλαδή ε, θα μετακινήσει διάφορα μέτρα της εξωτερικής πολιτικής σε μία περίοδο επταετίας αυτό τι συνεπάγεται από πλευράς μειώσεων των αμέσων εκλεξίμων δαπανών της Ευρώπης για την ε, αναπτυξιακή βοήθημα και σε περίπτωση που ε, επικροτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι προτάσεις αυτές μπορούμε να εξασφαλίσουμε η τα ποσά αυτά που θα αφαιρεθούν από το DCI και θα χρησιμοποιηθούν στο έρασμους μούντους να παραμείνουν επιλέξιμες, ε, επιλέξιμα τα ποσά αυτά ως αναπτυξιακή βοήθεια. Δηλαδή, εάν δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την πρόταση αυτή, θα ήθελα να ξέρω εάν μπορούν να ανατεθούν αυτές ε, οι να χρησιμοποιηθούν αυτά τα ποσά για να προωθήσουν τους στόχους τους οποίους έχουμε καταρτήσει. Ο Φελίξ. Φίλιξ, μάλλον. Αλλά όχι, προηγουμένως. Θέλεις να, θέλει κάποιος να απαντήσει στην ερώτηση του Τσάρλς. Νομίζω ο Φιλίπ. Νομίζω ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι η χρηματοδότηση του DCI έχει κάποια δυνατότητα προσαρμογής και Νομίζω ότι το άρθρο που αναφέρεται στο Erasmus Mundus λέγεται ότι θα περιληφθεί ε, στις προτεραιότητες του DCI και άρα στις ε, ανάγκες του DCI. Δηλαδή δεν θα υπάρχει μεταξύ μετακίνηση από το DCI κάπου αλλού για να εξυπηρετηθεί το Erasmus Mundus. Υπάρχει η νόμιμη προϋπόθεση τα χρήματα του DCI να διπλασιαστούν. Και αυτό νομίζω είναι αυτό το οποίο προβλέπουμε. Αυτό είναι και το πρόβλημά μας, λέει ο Πρόεδρος. Ο Τσάρλς θα ήθελε να αλλάξουμε την κατάσταση αυτή. Πώς θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις προοπτικές. Ο κύριος Γκάρενς έθεσα δύο ερωτήσεις. Μετά θα κάνω τα σχόλια και τις κρίσεις. Προς το παρόν ρώτησα. Σύμφωνα με ποιες διατυπώσεις ε, το, τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν. Δηλαδή αν λέγεται έρασμους μούντους δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβάλλει στην ε, ανάπτυξη του DCE. Αλλά αυτό θα το δούμε όταν θα εξετάσουμε την κοινοβουλευτικά έγγραφα. Ε, ο, απάντηση από την Επιτροπή. Ε, νομίζουμε ότι συντάσσουμε διάφορα προγράμματα τα οποία υπάρχουν ήδη και, τα και συγκροτούμε ένα σύνολο. Υπήρχε κατακαιρματισμός και η ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να συγκεντρωθούν μόνο υπό μία επικεφαλίδα όλα τα χρήματα αυτά με δύο πηγές χρηματοδοτήσεως στο κεφάλι κεφάλαιο 1 και στο κεφάλαιο 4. Και στο κεφάλαιο 4 θα χρηματοδοτηθούν μέσω των διαφόρων γεωγραφικών μέτρων συμπεριλαμβανομένων και του μέτρου για τις συνεργασίες. Εάν ε, υπάρχει μεταφορά ερευνητών από τις τρίτες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις δυνατότητες των συνεργαζομένων ε, κρατών σε πλαίσια του έρασμους μούντους ε, θα υπάρχει πλήρη κάλυψη και θα μπορέσουμε να καλύψουμε κατά αυτόν τον τρόπο την μετακίνηση Ευρωπαϊκή Ευρωπαίων φοιτητών προς τις χώρες και άπαξ και προκύψει η υποχρέωση βάσει των ε, γεωγραφικών προγραμμάτων να υπάρχει μία κάλυψη κατά 100% για να ε, υπάρξει αυτή η κάλυψη δεν θα μπορέσει πλέον να ε, ε, χρηματοδοτηθεί η κινητικότητα των φοιτητών προς τις τρίτες χώρες από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια αυτού του συνόλου. Και αυτό για να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα προτείνουμε μέτρα τα οποία δεν θα συνάδουν με τους κανόνες του ΟΣΑ. Δεν έχουμε χρόνο. Ο Φίλιπ να, συ... να συνεχίσεις αυτά τα οποία έλεγες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ενδεχομένως νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε με ό,τι είπε ο εισηγητής στα οικονομικά θέματα. Έχουμε πλήρη συνείδηση και θέλουμε να προστατεύσουμε ακριβώς για τους λόγους που είπατε την ε, χρηματοδότηση της ανάπτυξης όχι μόνο στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αλλά και στα κράτη-μέλη και εγώ θα επικεντρωθώ σε δύο-τρία σημαντικά θέματα εκ των οποίων το πρώτο είναι ότι αυτό είναι μία εφαρμογή ε, που αντικατοπτρίζει τις ε, τη συζήτηση που είχαμε, την Agenda for Change, με, σε νομικούς όρους. Και αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε είναι όχι μόνο τις προτεραιότητες, αλλά όπως είπατε και εσείς, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειάζεται ένας ρυθμιστικός κανονισμός που να καλύπτει τις προϋποθέσεις τις οποίες ζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και από τη μία πλευρά υπάρχει προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα διότι όπως ελέγχθη προηγουμένως πρέπει να προωθήσουμε όλο και περισσότερο το γεγονός για να προβάλλουμε ότι τα κράτη-μέλη θέλουν να περάσουν ένα μήνυμα προς τους εταίρους μας όλοι μαζί για να έχει μεγαλύτερο βάρος αυτό το μήνυμα και έχουμε να στείλουμε ε, πολλά σημαντικά μηνύματα όχι μόνο ως πολιτικά μηνύματα αλλά ε, και με εφαρμογή των μηνυμάτων στην πράξη. Και ένα από αυτά τα μηνύματα είναι πώς θα εξηγήσουμε και θα στηρίξουμε τις υποανάπτυξη χώρες για να προωθήσουν διάφορα θέματα που ανέφερε ο εισηγητής μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Χρειαζόμαστε ε, παρκές βάρος για να μπορέσουμε ε, να προβάλλουμε τα θέματα αυτά σε συζητήσεις και γενικότερες και μεταξύ μεμονωμένων κρατών για να περάσει το μήνυμα ευκρινώς και ε, φαντάζομαι ότι αυτό το καταλαβαίνετε. Και με αυτά πανερχόμαστε στην πολιτική της διαφοροποίησης διότι η διαφοροποίηση είναι μία πολύ θαραλέα πρόταση και ενδεχομένως ε, ορισμένοι μπορεί να κατακρίνουν την ε, απλότητα της προτάσεως αλλά πρέπει να δούμε και το αποτέλεσμα αυτής της απλότητας και αντιλαμβάνεστε ότι ε, υπάρχουν χώρες όπου υπάρχουν οι περισσότεροι φτωχοί άνθρωποι στον κόσμο και πρέπει συγχρονώς να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχει προστιθέμενη αξία και επίπτωση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην μείωση της φτώχειας. Υπάρχουν ε, πολλές φτωχές ε, χώρες και πολλές χώρες μέσου εισοδήματος και όπως είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε ε, το κριτήριο που θα είναι το πιο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να επιλύσουμε τα προβλήματά τους στις στόχες ή να τους υποκινήσουμε ε, πολιτικά να το πράξουν και ε, εάν υπάρχει μικρή εξάρτηση μπορούμε να, χρησιμο... να θεωρήσουμε ότι ορισμένα από τα χρήματα που θα αφιερώναμε εκεί θα είναι πιο αποδοτικά κάπου αλλού δηλαδή στις, ε, μέσω, στις ε, χώρες μέσου εισοδήματος μήπως θα έπρεπε να μετατεθούν στις στοχότερες χώρες για να υπάρχει μία πιο σημαντική προβολή και αυτό είναι μια πολιτική απόφαση που πρέπει να ληφθεί και είναι στο χέρι σας και στο χέρι του Συμβουλίου εάν θα συνενέσει σε μια τέτοια λύση και πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση και θα σταματήσω σε αυτό το σημείο. Ευχαριστώ Φίλιξ. Θέλω να επανέλθω στο θέμα αυτό. Ε, ε, όλα αυτά βέβαια προϋποθέτουν ότι οι χώρες μέσου ε, οικονομικού επίπεδου έχουν τη δυνατότητα να λύσουν τα προβλήματα των φτωχών συνοικιών και να προωθήσουν την ανάπτυξη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη εάν μιλάμε για την Κίνα θα μας πούν μην έρχεστε στη Σανγκάη και στις ε, περιοχές ε, που είναι κοντά στη θάλασσα αλλά ελάτε στο εσωτερικό της χώρας να δείτε τι γίνεται όπου δίπλα στους ε, μεγάλους ουρανοξύστες υπάρχουν παράγγες και δημιουργήστε την θέληση να εξαλειφθούν αυτές οι παράγγες και θέλω να χαιρετήσω τώρα τον εκπρόσωπο της ε, Προεδρίας του Συμβουλίου και βλέπω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου θα συμμετάσχει στη συζήτηση και ζητώ από τον κύριο Νίκολς να λάβει τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που με έχετε προσκαλέσει ως Πρόεδρο του Σώματος Εργασίας ε, για την Αναπτυξιακή Συνεργασία να σας παρουσιάσω την κατάσταση ε, στην ομάδα εργασίας ε, σε σχέση με το TCI. Τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν μια σε βάθος ανάλυση της πρότασης που όπως φαντάζεστε απαιτεί χρόνο και προσοχή. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέπεια και συνεκτικότητα όλων των μέσων ε, εξωτερικής ε, δράσης και διάστασης. Γι' αυτό χρειάζεται στενή συνεργασία και με τις άλλες ομάδες εργασίας. αλλά και με την ομάδα εργασίας φίλη της Προεδρίας σε σχέση με τον εφαρμοστικό κανονισμό και τα οριζόντια ζητήματα. Σε σχέση τώρα με την κατάσταση, ένα βασικό μήνυμα είναι ότι η Ιδανική Προεδρία έχει ως συνολικό στόχο μια γενική συμφωνία για όλα τα μέσα μέχρι τα τέλη Ιουνίου, ε, υπό, την, ε, υπό μια ενιαία δέσμη. Αυτό είναι το χρονοδιαγραμμά μας. Το του λεχθέντος πρέπει να προσθέσω ότι τα βασικά στοιχεία της θέσης του Συμβουλίου βρίσκονται σε πολύ προκαταρκτικό στάδιο ακόμα. Θα σας αναφέρω δύο-τρία από αυτά με πάρα πολλές επιφυλάξεις και περιορισμούς μέχρι στιγμής. Το Συμβούλιο φυσικά επιθυμεί να υπάρχει ε, ο συμβασμός ιδίως ό,τι αφορά την ατζέντα για αλλαγή και πάνω σε αυτό να οικοδομήσει. Το Συμβούλιο χαιρετίζει την καινοτόμο προσέγγιση που προτείνεται για το μέσο εξωτερική βοήθεια και υποστηρίζει πλήρω την ιδέα να εστιάσει περισσότερο σε αυτό και να υπάρχει και μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Χαιρετίζουμε επίσης την ευελιξία και την ανταπόκριση που υπάρχει, αλλά πρέπει να δούμε με ποιον τρόπο θα πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Η Προεδρία είναι αισιόδοξη ότι θα είναι επικοδομητικέ συζητήσει στο Κοινοβούλιο και θα εξασφαλίσουν ε, την ε, έγκαιρη υιοθέτηση αυτών των μηχανισμών για να υπάρχει συνέχεια στην εξωτερική δράση τη Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ κύριε Νίκο. Δεν ξέρετε πόσο ευγνώμων σας είμαι που ήρθατε εδώ να μας πείτε αυτά πολύ σημαντικά που μας είπατε. Θα σας δώσω τώρα κύριε Μπέρμαν σε εσάς το λόγο για να καταλήξετε πολύ σύντομα. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν με επιτρέπετε, επειδή έχει πέρασει ο χρόνος... Ναι, έχει πέρασει ο χρόνος, λίγε παρατηρήσει μόνο. Αυτό που είπε ο Ρικάρντο και για την έκθεσή του στην Επιτροπή ΑΦΕΤ. Θα έχουμε το σχέδιο έκθεση έτοιμο τον επόμενο μήνα και θα γνωμοδοτήσουμε η Επιτροπή ΝΤΕΒ από αυτού του σχεδίου έκθεση και θα πρέπει και με την ΑΦΕΤ για τα οριζόντια στήματα να συντονιστούμε για να υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ των δύο εκθέσεων για την προσέγγιση βάση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα ήθελα να πω ότι τελικά, ακόμη και αν υπάρχουν κείμενα στην πρόταση για τον DCI, πολύ σωστά μιλήσατε για το άρθρο 3.1, αλλά και για το τελευταίο άρθρο και στην πρόταση που λέει ότι εάν οι χώρε εταίροι δεν πληρούν τις υποχρεώσεις του ό,τι αφορά σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτος δικαίου, θα μπορούσε να ανασταλεί η βοήθεια. Ναι, ναι, ναι, αλλά ένα είναι το ερώτημα. Έχει την πολιτική βούληση Ευρωπαϊκή Ένωση. Να είναι δηλαδή μια ένωση με το πολιτικό της βάρος, ε, με την βούλησή της, της αξίας της και μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη βάσει των δικαιωμάτων των πολιτών και στο πλαίσιο βιώσιμης ανάπτυξης έχει αυτή τη φιλοδοξία η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια δεν είναι μόνο η Κομισιόν και τα κράτη-μέλη και το Κοινοβούλιο πρέπει να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Θα ήθελα να επιδείξει πολύ μεγαλύτερη φιλοδοξία και πολύ πιο ξεκάθαρα να αναφέρει αυτούς τους στόχους και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί το λένε και τα νομικά μας κείμενα. Αυτό. Για τον Γκέι κάτι τελευταίο. Πολλά καλά είπε. Ο ε, πρέπει πράγματι να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν ε, πάρα πολλά κοινά στοιχεία Μίλησες και για το πρόβλημα του φύλου, ε, για τους στοχούς πληθυσμούς και για κάποιες ε, άλλες ε, ομάδες, ότι έχουμε πάρα πολλές αμβλώσεις, ιδίως όταν είναι το έμβριο θηλυκού γένους. Πράγματι, όλα αυτά μπορούν να περάσουν τρομερά τη ζωή των πληθυσμών και ίσως πράγματι και εμείς έχουμε να διαδραματίσουμε ένα πολιτικό ρόλο. Γιατί δεν πρέπει να ενισχυθούν μόνο τα οικονομικά δικαιώματα. Πρέπει να προωθήσουμε τα ίσα δικαιώματα για τους άνδρες και τις γυναίκες. Γιατί έτσι θα αλλάξει και αυτή η εικόνα άρδιν. Και θα σταματήσω με αυτό το σχόλιο. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Τέις. Θα συνεχιστεί η συζήτηση για το νομοθέτημα αυτό. Και τώρα πάρα πολύ γρήγορα πρέπει να ασχοληθούμε με ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα, τις άμεσες ε, πληρωμές. στι πληρωμέ υπέρ των γεωργών στο πλαίσιο του καθόλου στήριξη, κοινή οργάνωση των αγορών γεωργικών προϊόντων, στήριξη αγροτική ανάπτυξη, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτική Ανάπτυξη κτλ. Έχουμε τον αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή τη ε, ΑΜΚΟ εδώ, αλλά δυστυχώς ε, πρέπει να φύγει σύντομα και η κυρία Σνίμπερ Γιάστρα, μην συγκίτριά μας. Θα ζητήσω από την συγκίτρια να Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα για την Επιτροπή Ανάπτυξης που είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό λυπάμαι πάρα πολύ ότι πρόκειται τώρα να το συζητήσουμε με τόσο, σε τόσο περιορισμένο χρόνο. Θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομη και να αναφερθώ μόνο σε ορισμένα θέματα και να ευχαριστήσω τον Γιάννη και για την στήριξή του. Έχουμε επενδύσει πάρα πολύ χρόνο σε αυτό το τομέα που είναι ένα πολύ βασικό θέμα και θα μπορούσε πολιτικά να είναι τελείως διαφορετική αυτή η μεταρρύθμιση, πιο φιλόδοξη, ε, πιο εστιασμένη ε, όσον αφορά τις αποδεσμευμένες πληρωμές. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχουν και πολλές ασυνέπειες ε, στο παρελθόν οι οποίες μετά διορθώθηκαν και πιστεύουμε ότι είμαστε στη σωστή οδό όσον αφορά την πράσινη ανάπτυξη που ανέφερε ο Επίτροπος και ε, υπάρχουν και άλλες δυνατότητες να προωθήσουμε το θέμα της έρευνας και της ανάπτυξης που είναι σημαντικό και για τις δύο πλευρές και για τη γεωργία και για την αναπτυξιακή βοήθεια. Σε όλους τους τομείς έχουμε συζητήσει ότι είναι βασικό να είμαστε συνεκτικοί και συνεπείς ε, με την ε, ε, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως γιατί βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που πολλοί δεν αντιλαμβάνονται πόσο σημαντικό είναι αυτό. Δεν έχουμε τοποθετηθεί, μάλλον δεν έχουμε τοποθετηθεί διαφορετικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις ποσοστώσεις της Ζαχάρεως η οποία εκπνέει και η Ευρωπαϊκή και η Επιτροπή μας έχει διαφορετική αντίληψη αλλά θα το εξετάσουμε στη συνέχεια. Επίσης οι ποσοστώσεις πρέπει να σταματήσουν στο τέλος του 2017. Υπάρχουν δηλαδή διάφορες τροπολογίες οι οποίες θα υπάρξουν και εγώ δεν θέλω να επιβαρύνω υπερβολικά το κείμενο διότι θα υπάρχει δυσκολία να συντονιστούμε με τους υπευθύνους για τη γεωργία. Είμαστε όμως σε καλό δρόμο, δεν έχω ακούσει κραυγές εκπλήξεως και τρόμου και πιστεύω ότι έχουμε πετύχει πολλά περισσότερα σε αυτή την ε, γενικά ενιαία αντιμετώπιση. Δηλαδή ε, πρέπει να είναι σαφές ότι δεν ζητούμε μια αντιπαράθεση αλλά προσπαθούμε όλοι μαζί να ακολουθήσουμε το σωστή οδό. Θα μπορούσα να σας πω πολύ περισσότερα, τώρα θα περιοριστώ, προσβλέπω στις συζητήσεις, ε, στα σχόλιά σας, έχω χρόνο διαθέσιμο και σας παρακαλώ να μην επιβαρύνουμε υπερβολικά την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Εδώ πρωτοπορούμε θα έλεγα. Διότι έχει πλέον ε, δυνατότητες συναπόφασης, αρμοδιότητες συναπόφασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ακόμα και σε σχέση με την ΚΑΠ. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία, την οποία θα χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι ώστε να βελτιώσουμε την κατάσταση αυτή. Θα ξεκινήσει η συζήτηση τώρα με τους συναδέλφους. Ο Ρικάρντο. Θα ήθελα εγώ να ευχαριστήσω την κυρία Χάστρομ για την εξαιρετική δουλειά και την προετοιμασία των γνωμοδοτήσεων αυτών. Στηρίζει πλήρω η ομάδα μα και πρέπει να είναι συνεκτικές προσπάθειε της Ένωσης στην αναπτυξιακή συνεργασία. Στηρίζουμε επίσης ε, και τις μελέτε αντικτύπου τη κοινωνική πολιτική. και ελπίζουμε η Επιτροπή Άγκρη να εγκρίνει την πολύ σημαντική σχετική πρόταση. Η δική μας ομάδα πάντοτε ήταν αντίθετο με τις επιδοτήσεις της ε, εξαγωγές. Γι' αυτό συμφωνούμε απόλυτα με την πρόταση να δοθεί ένα τέλος σε αυτού του είδους τις επιδοτήσεις. Ένας από τους στόχους μας και θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να αποσυνδεθούν ε, οι ενισχύσεις για την πολιτική και θα πρέπει να καταργηθεί η, στρέβλωση που υπάρχει, το trade distortion, οι εμπορικές διαστρεβλώσεις. Στηρίζουμε επίσης τις προτάσεις που σχετίζονται με την επιστημονική έρευνα προς όφελος των ψώμενων χωρών. Uh, Ευχαριστώ, Ρικάρντο. Κριστίνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, συντάκτρια και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε γιατί συμφωνώ ότι είναι ένα βασικό θέμα δηλαδή η διασύνδεση της γεωργίας με την αναπτυξιακή προοπτική καθότι ε, θα έχουμε μία πληθυσμιακή έκρηξη ανθρώπων που δεν θα ζουν στην Ευρώπη αλλά στις υποανάπτυξη και αναδυόμενες χώρες θα με περισσότερη παραγωγή και θα χρειαζόμαστε να έχουν δυνατότητες προωθήσεως και τα προϊόντα που παράγονται επί τόπου. Ε, και παραδείγματος ε, χάλι να ε, πρέπει να θυμηθούμε ότι στο δέλτα του Νείλου μπόρεσαν να προωθηθούν παρόλου του υφάλα του ύδατος καλλιέργειες οι οποίες ήταν πολύ αποδοτικές και ε, όλες αυτές οι επιδοτήσεις ε, ε, ουσιαστικά για την Ευρώπη είναι ένα μικρό ποσό και καλό θα ήταν να μπορέσουμε να τις εξαλείψουμε. Βέβαια η Ευρώπη είχε πολύ καλή θέση για τα τρόφιμα και την πρόθεσή τους στην Ευρώπη και όταν συγκρίνουμε με άλλες περιοχές περιοχές όπως ε, η Νέα Ζηλανδία θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα προωθήσουμε τα συμφέροντα της Ευρώπης αλλά νομίζω ότι μπορώ να στηρίξω αυτά τα οποία είπατε προηγουμένως. And, uh, Ο κύριος Πατσέκο, αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής ε, στην Γεωργία, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω κάτι το οποίο είδα στην πρότασή σας, ότι οι προτάσεις μας ε, για την μεταρρύθμιση της ΚΑΠ ακολουθούν, θα έλεγα, αυτά τα οποία έχετε ζητήσει εσείς τα τελευταία δέκα χρόνια έτσι ώστε να μην υπάρξουν στρεβλώσεις στο ε, εμπόριο. Υπάρχουν, ε, υπάρχει άμεση βοήθεια η οποία δεν προκαλεί αρνητικές επιπτώσεις στις υπόλοιπες χώρες. Έχουμε έτσι και αλλιώ εκ των υστέρων αξιολογήσεις στις πολιτικές μας, δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις και προσπαθούμε να εξετάσουμε επίσης και τις επιπτώσεις της πολιτικής μας σε όλες τις υπόλοιπες πολιτικές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα τον τομέα των αναπτυξιακό. Για τα συγκεκριμένα θέματα στην έρευνα και στην ανάπτυξη, εμείς προτείναμε ένα τεράστιο βήμα προς τα εμπρός σε επίπεδο πόρων, θεωρούμε και ελπίζουμε να μας υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και είμαι πεπισμένος ότι η έρευνα και η ανάπτυξη που κάνουμε θα ωφελήσει και τις αναπτυσσόμενες χώρες. Κατανοώ επίσης τις θέσεις σας στον τομέα των εξαγωγών. Καταρχάς, έχουμε προγραμματίσει τις επιστροφές στις εξαγωγές να τις ε, εξαφανίσουμε σε εισαγωγικά σταδιακά και είχαμε πει ότι όταν είχε κλείσει ο γύρος της Ντόχα θα είχαμε τελειώσει με τις επιδοτήσεις εξαγωγές αλλά δυστυχώς ο, ο γύρος της Ντόχα συνεχίζεται ακόμα και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο μονομερός γιατί εμείς θέλουμε κάποιοι καλύτεροι μηχανισμοί για την υποστήριξη των εξαγωγών από άλλες αναπτυχόμενες χώρες να καταργηθούν και αυτοί. Ως εκ τούτου λοιπόν θα πρέπει να συνεχίσουμε να παίζουμε με αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί. Βέβαια η παρούσα κατάσταση δείχνει ότι όχι μόνο το 95% των δαπανών μας πηγαίνει σε επιστροφές στις εξαγωγές, αλλά από τις δαπάνες αυτές μόνο το 10% χρησιμοποιείται για χώρες οι οποίες ταξινομούνται σαν αναπτυσσόμενες. Και πρέπει να πω με μεγάλη ικανοποίηση ότι την προηγούμενη εβδομάδα εμείς για ορισμένα προϊόντα είχαμε μηδενικές επιδοτήσεις και έχουμε ε, για κάποια προϊόντα για την Ιαπωνία μόνο, Σαουδική Αραβία, ε, η και ιδιαίτερα ε, σε τομείς όπως η παραγωγή κρέατος ε, που είναι τελικά περιθωριακό στο σύνολό μας. Λοιπόν, δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο άλλο σχόλιο. Πριν δώσω το λόγο ξανά στην κυρία Άιστρομ. Δεν θέλω να παρατείνω τη συζήτηση. Ευχαριστώ για τις τοποθετήσεις και ε, θα το ξανασυζητήσουμε όταν θα υπάρξουν άλλες απαιτήσει και θα δούμε. Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για μας τίθεται το θέμα ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο γύρος της Ντόχα και αναρωτιόμαστε εάν δεν θα έπρεπε και σαν Επιτροπή Ανάπτυξης να θέσουμε το ίδιο ερώτημα και την ίδια απέτηση με επιτρέπετε για 27 λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Είχαμε τη γαλακτοκομική κρίση πριν από κάποια χρόνια και έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σταθεροποίηση των τιμών τα κονδύλια της τιμής του γάλακτος. Δεν θα ήθελα να ξανα... Τέλος πάντων δεν το βλέπω να ξανασυμβαίνει. Thank you very much. Ευχαριστώ. Θέλετε να απαντήσετε. Κατάλαβα τι λέτε. Εμείς δεν χρησιμοποιούμε για τα γαλακτοκομικά προϊόντα επιστροφή, επιστροφή ε, εξαγωγών. Δεν προβλέπουμε να χρησιμοποιηθεί λοιπόν στο μέλλον άμεσα τουλάχιστον ο μηχανισμός αυτός. Κάποιος άλλος. Όχι, άρα σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ζητώ συγγνώμη που το πήγαμε λίγο γρήγορα, αλλά τουλάχιστον δεκπεραιώθηκε το θέμα αυτό. Επόμενο. Η κοινή οργάνωση των αγορών και οργικών προϊόντων ε, και υπάρχει Έχουμε το την αξιολόγηση του αναπτυξιακού προγράμματος Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής από στην Επιτροπή Αναπτυξιακή Βοηθείας του ΟΣΑ και θα καλέσουμε τον πρόεδρο της Επιτροπής Αναπτυξιακή Βοηθείας ε, να έρθει στο Προεδρείο για να το συζητήσουμε από κοινού. Um, the timing of Mr. Atwood's visit coincides with the official launch of the DAC. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η αξιολόγηση ομοτήμων τη ΔΑΚ, ε, του ανθρωπιστικού προγράμματο, ανθρωπιστική βοήθεια τη Ένωση, ε, και με αυτό συμπίπτει η παρουσία του κ. Μπράιαν Άτχουτ. Σήμερα, πολύ επίκαιρα έχουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχουμε την μοναδική δυνατότητα να συζητήσουμε για πόλεμο τον κύριο Άτχουτ τι βασικέ συστάσει της ΝΤΑΚ για την ιδιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ακούσουμε και την αντίδραση της Κομισιόν. Τελική έκθεση της αξιολόγησης ομοτήμων έχει, δια, έχει διανεμηθεί. Στόχος του ΝΤΑΚ είναι η πρόθεση των βέλτιστων πρακτικών, συνεργασίας. Πάντα ήταν ένα σημείο αναφοράς, πολύ σημαντικό. Συζητήσαμε σήμερα το 20% για την υγεία, την εκπαίδευση, Η ΔΕΒ έχει βασιστεί πολύ και στο έργο της ΔΑκ Ο ΣΑ δημοσίευσε ένα πολύ σημαντικό έγγραφο πρόσφατα που δείχνει σχετικές τάσεις. Δηλαδή, αντί να έχουμε το 0,7% για την αναπτυξιακή βοήθεια, το 11 τα 27 κράτη-μέλη απομακρύνθηκαν από το στόχο αυτό. 0,42 από το 044 στο 10. Και γι' αυτό θα πρέπει να ξέρουμε ότι ναι μεν δεν είναι η ποσότητα το παν για την αψυχή βοήθεια, αλλά και η ποιότητα. Και εκεί θα επικεντρωθούμε σήμερα. Θα δώσω στον κύριο Άτκου το λόγο για να μας παρουσιάσει την αξιολόγηση των Αναπτύξου προγράμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Επιτροπή Αναψυχίας Βοήθειας ΔΑΚ του ΟΣΑ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να σας πω ότι είναι τιμή για μένα που βρίσκομαι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα προσπαθήσω να μην παρέμβω στην νομοθετική διαδικασία μετά όσα θα πω. Θα προσπαθήσω αντικειμενικά να σας μεταφέρω την αξιολόγηση από ομοτήμους και το τι μας λέει. Μία αξιολόγηση η οποία έγινε από δύο άλλες χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ιαπωνία και η Νορβηγία και η διαδικασία ήταν μία ε, αποστολή στις Βρυξέλλες για μία εβδομάδα, τον Οκτώβριο, και επιστροφή εδώ ε, το Δεκέμβριο και είχαμε και συνεδριάσεις με μη κυβερνητικέ οργανώσεις, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και με βουλευτές. Νομίζω ότι ήταν μια ενδελεχής διεξοδική διαδικασία. Δύο επισκέψεις πραγματοποιήθηκαν σε δύο χώρες όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εξέχουσα παρουσία. Τσάντ στην Αφρική και Περού στη Λατινική Αμερική. Δύο πολύ διαφορετικές χώρες, η μία μεσαίου εισοδήματος και η άλλη πολύ χαμηλού εισοδήματος. Χώρα με πολύ εύθραυστο κράτος. Καταρχάς θα ήθελα να σας αναφέρω το πλαίσιο. Είναι πολύ σαφή η μοναδικότητα ε, της δράσης Ευρωπαϊκής Ένωσης που βέβαια μοιάζει πολύ με μια διμερή ε, οργάνωση παροχής βοήθειας ο τρόπο με τον οποίο εργάζεται η Κομισιόν, αλλά από άλλε ενίες είναι πολυμερή η προσέγγιση γιατί υπάρχουν υπάρχει συμμετοχή από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Πίτροπος Πίλμπαξ λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα sui generis μέλος ε, της ε, ΔΑΚ, της Επιτροπής Αναπτυξικής Βοήθειας του ΩΣΑ. Τι κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι το πλαίσιο των επιχειρήσεων. Είναι η συνθήκη της Λισαβόνας φυσικά, η οποία βέβαια διέπει τις μάλλον τις ε, δράσεις αναπτυξιακής συνεργασίας της Ένωσης ε, με μεγάλες αλλαγές. Ένας στόχος της συνθήκης ήταν μεγαλύτερη συνεκτικότητα της εξωτερικής πολιτικής της Ένωσης. Ένα πολύπλοκο λοιπόν θεσμικό και ε, ένα πολύ πολύπλοκο θεσμικό σύστημα το οποίο ήταν η απόρρια της συνθήκης. Και πρέπει να σας πω επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει και έναν ρόλο ομοσπονδοποίηση κατά κάποιο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά έχει διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της αναπτυξιακής κοινότητας. 70 δις δολάρια από 130 δις που παρέχει, δηλαδή πάνω από το 50% και στο βαθμό που παίζει αυτόν τον ρόλο, τον ενωτικό, ε, συνάδει αυτό ο ρόλο με τον ρόλο που προσπαθούμε και εμεί στην Επιτροπή Αναπτυξιακή Συνεργασία να διαδραματίσουμε. Ένα σημαντικό λοιπόν εταίρο τη ΔΑΚ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω σα είπα, ε, και άλλωστε και το 50%, πάνω από το 50% των μελών τη ΔΑΚ είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεργαζόμαστε στενά λοιπόν και ήταν πάρα πολύ ενθαρρυντικό και βοήθησε την όλη διαδικασία αυτή η ατζέντα για την αλλαγή που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο πριν την συνεδρία στην Κορέα, στο πουσά Για τη συνεργασία, για την αναπτυξιακή συνεργασία. Εμείς συμφωνούμε πλήρως με το όραμα της ατζέντα για την αλλαγή. Γνωρίζουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μελετά το όλο θέμα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών διευθετήσεων. Είναι πολύ έγκυρη η στρατηγική αυτή αντίληψη και στο Μπουσάν είχε ασκήσει ιδιαίτερη επιρροχή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο στοιχείο είναι το παγκόσμιο πλαίσιο, το γενικότερο πλαίσιο. Θα ήθελα να σα πω τι συνέβη στο Μπουσάν, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό. Στο Μπουσάν οι αναπτυσσόμενε χώρε ουσιαστικά πήραν ε, τα ενία. Αυτό ήταν το σημαντικότερο ε, στοιχείο. Είχαμε πολλά φόρουμ ψηλού επίπεδου που τα μέλη τη ε, ΝΤΑΚ και στην δήλωση των ε, Παρισίων όπου θέσαμε κάποιες αρχές ε, και γενικώ είχαν τα ενία. Αυτή τη στιγμή όμως είμαστε πιο ταπεινοί πηγαίνοντας στον Μπουσάν γιατί με κάποιες έρευνες ε, που κάναμε είδαμε ότι έναν από τους 13 μόνο στόχους που είχαμε ορίσει ε, μέσω της διακήρυξης των Παρισίων είχαμε εφαρμόσει τελικά. Και με βάση την αξιολόγηση που κάναμε πιστεύουμε ότι είναι σωστές οι αρχές αυτές για τη δημιουργία, για την επιτυχία επίτευξη ανάπτυξης, αλλά δεν τα καταφέραμε πολύ καλά, δεν κάναμε πολύ καλή δουλειά. Θέλαμε λοιπόν οι αναπτυσσόμενε χώρε να είναι αυτέ οι οποίε θα πάρουν τα ενία όπω και έπραξαν. Και το σημαντικότερο μήνυμα στον Μπουσάν είναι ότι πρέπει να προσέξουμε την ιδιοκτησία, ε, την οικειοποίηση δηλαδή του προγράμματος από την εκάστοτε χώρα. Είδαμε σημαντικές βελτιώσεις στα στατιστικά συστήματα κτλ. Είδαμε βελτίωση κατά 33%. Μόνο το 8% της αναπτυξικής, επίσημης αναπτυξικής βοήθειας είχε περάσει μέσα από αυτά τα συστήματα. Οι αναψώμενες χώρες λοιπόν είχαν πρόσβαση σε όλες αυτές τις πληροφορίες και για κάποια πράγματα πίεσαν όπως ε, για τις αρχές ε, του Παρισιού, προβλεψιμότητα κτλ. Η διάσκεψη του Μπουσάν είναι πολύ σημαντική και έχει να κάνει αυτό με τις δικές σας ε, ανησυχίες για τον προπολογισμό, τις γενικές κατευθύνσεις που παρέχετε προς την Κομισιόν για αυτά τα θέματα. Ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε το ότι περνάμε από μία σχέση συναλλαγών σε μία σχέση αναπτυξιακής αποτελεσματικότητας. Πάρα πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει συνεκτικότητα στην πολιτική εσείς έχετε αναλάβει δεσμεύσει, έχετε σε αυτά τα θέματα, να υπάρχει συνεκτικότητα στις πολιτικές. Νομίζω ότι και εμείς τονίσαμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έναν ηγετικό ρόλο ε, στην συνεκτικότητα της πολιτικής, αλλά η υλοποίηση των σχετικών δεσμεύσεων ε, δεν είναι ομοιόμορφη από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Είδαμε λοιπόν τις επιδόσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί δεν είναι μόνο τι κάνει και τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι αν σας δίνουν τα κράτη-μέλη την πολιτική ε, βούληση για να κάνετε τα λόγια έργα. Υπάρχει μια πολύ σημαντική αρχή λοιπόν, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά γενικότερα, ε, τα κράτη που χρηματοδοτούν ε, δεν έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά έχουμε ουσιαστικά υπονομεύσει με πολιτικές εγχώριες ε, τις επενδύσεις. Αφαιρούμε κίνητρα, παραδείγματο χάρη, για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα κτλ. Στην ατζέντα για την αλλαγή αλλά και στη συμφωνία του Μπουσάν περιλαμβανόταν ε, η εργασία με εύθραυστα κράτη Είχαμε κάποιες συναντήσεις στην Ουάσιγκτον, ήταν και κάποιοι από τους υπουργού σας παρόντες, έγινε συζήτηση εκεί για το νέο deal, τη νέα συμφωνία που επιτέχθη στο Μπουσάν με τα έφραυστα κράτη, τα ευάλωτα κράτη, που από μόνα τους, είναι σημαντικό αυτό, έλαβαν την ευθύνη για το τι θα πράξουν για να έχουν την ίδια ιδιοκτησία και την, να αγκαιοποιηθούν τα προγράμματά τους. Και Κάποιες ευρωπαϊκές χώρες επίσης δεσμεύτηκαν σε περιοχές υψηλού κινδύνου να αναλάβουν δράση. Είναι σημαντικό λοιπόν να παρασχεθεί απαραίτητη υποστήριξη ώστε να συνεχιστεί αυτό το έργο. τα αποτελέσματα τα οποία μπορούν να επιτευχθούν σε χώρε μεσαίου εισοδήματο ή σε πολύ σταθερότερε χώρε ε, ε, δεν θα επιτευχθούν σε αυτέ τι ευάλωτε ή έφραστε χώρε, αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να επενδύσουμε στι χώρε αυτέ, γιατί αν δεν καταφέρουν να σταθεροποιηθούν, τότε θα χρειαστεί να έχουμε στρατιωτικέ δυνάμει, ενευτικέ δυνάμει, ανθρωπιστική βοήθεια από τα Ηνωμένα Έθνη που θα πρέπει να πάει σε αυτέ τι κοινωνίε. σε αυτά τα κρατή. Άρα πάρα πολύ σημαντική αυτή η νέα συμφωνία και επίσης η κοινωνία των πολιτών και ο ιδιωτικό τομέα συμμετείχαν στη συμφωνία του Μπουσάν και συμμετέχουν στην ατζέντα για την αλλαγή. Όταν λέμε ότι θέλουμε οι χώρες να οικειοποιηθούν, να ιδιοποιηθούν τα προγράμματά τους, δεν μιλάμε για τις κυβερνήσεις μόνο, μιλάμε για τους πολίτες. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Ο πρόεδρος ανέφερε τα επίπεδα της επίσημης αντιστικής βοήθειας. Νομίζω ότι, όπως λέμε και εμείς στην έκθεσή μας, δεν ε, είστε σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων και την τήρηση των δεσμεύσεων που έχετε αναλάβει. Και αυτό είναι άκρο ε, ε, αξιοπερίεργο, γιατί έχουμε προβλήματα γενικότερα. Υπάρχει μεγάλη μείωση στα επίπεδα 2,7% λιγότερη. Και είναι σημαντικό αυτό γιατί ξέρουμε ότι ο πλανήτης πλήττεται από οικονομική ύφεση. Πρέπει να συνεχίσουμε να ασκούμε πίεση πρέπει αυτό το 0,7% αυτός ο στόχος να τηρηθεί εγκαίρως, αν αυτό βέβαια είναι δυνατόν. Πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει επίπτωση, αν μειωθεί δηλαδή, αν συνεχίσει να μειώνεται η αναπτυξιακή αυτό θα επηρεάσει ακόμη περισσότερα τις χώρες ε, με χαμηλό εισόδημα. Στην έκθεση μεταξύ άλλων επισημαίνουμε και αυτό ε, γίνεται ίσω πιο πολύπλοκο λόγω τη συνδεκής τη Λισαβόνα, είναι ότι οι διαδικασίε είναι πάρα πολύ δυσκίνητες. Χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο για να συμβεί κάτι επί τόπου. Και δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγο να μην διορθωθεί αυτό. Αν βρεθεί η ευαρέτη πολιτική βούληση, μπορεί κάτι να γίνει. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν έχει διατυπώσει συστάσει στην Επιτροπή σα για να βελτιωθεί και να εξορθολογιστεί η διαδικασία και ελπίζω να εξετάσετε τις προτάσεις της Κομισιόν. Βέβαια, ο Μαξ Βέμπερ πριν από 100 χρόνια τουλάχιστον είχε προειδοποιήσει για το τι μπορεί να κάνει η γραφειοκρατία στη δημοκρατία. Προειδοποιήσει εξακολουθούν να υπάρχουν. Εγώ νομίζω ότι εσείς είστε δημοκρατία, εσεί έχετε την ευθύνη να δώσετε στην Κομισιόν τη δυνατότητα να εξορθολογήσει τις διαδικασίες της και να είναι πολύ πιο αποτελεσματική για την παροχή βοήθειας. Μια τελευταία λέξη. Με τον Επίτροπο Πίλμπαξ ε, ήταν μεγάλη μου χαρά που συνεργάστηκα, όπως και με τον Επίτροπο Γεωργίευα. Το ευχαριστήθηκα πραγματικά. Νομίζω ότι έχετε ικανότατους επιτρόπους ε, που ηγούνται, που κάνουν ό,τι μπορούν για να παίξουν αυτόν τον ε, ρόλο τον ενωτικό. Στο Μπουσάν έγινε σημαντική πρόοδος για την κοινό προγραμματισμό ε, η Ένωση είχε σημαντική συνεισφορά, προσπαθεί να βοηθήσει στον επιτόπο συντονισμό. Μια από τι προκλήσει που αντιμετωπίζουν οι χώρε είναι ο κατεκρεματισμό. Δηλαδή, πάρα πολλά προγράμματα, πάρα πολλά ταμεία παρακαταθήκων, trust funds κτλ. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα με τι 27 χώρε μέλη να προσπαθήσει να συνενώσει όλα αυτά και να ε, συντονίσει όλα αυτά τα προγράμματα. Πιστεύω ότι στον Μπουσάν καταφέραμε να κάνουμε τους Κινέζους, τους Ινδούς, τους Βραζιλιάνους, τους Νοτιοαφρικανούς, ε, τις χώρες BRICS ε, να ε, προσυπογράψουν τις ίδιες αρχές, βέβαια εθελοντικά, και στο πλαίσιο της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης για μια αποτελεσματική αναπτυξιακή συνεργασία νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε έναν καλύτερο μηχανισμό συντονισμού, να έχουμε διάλογο να δούμε τι συμπληρωματικότητες υπάρχουν στην συνεργασία Βορρά-Νότου και Νότου-Νότου. Έχουμε αναλάβει αυτή τη δέσμευση, την έχουν αναλάβει και οι άλλε χώρε και νομίζουμε ότι θα βοηθήσει τον επιμερισμό των βαρών, θα βοηθήσει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία επιτόπου και θα βοηθήσει κάποιε από ε, τι ε, απώλειες που είχαμε να τις ε, εξαλείψουμε. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά Ήμουν ο επικεφαλής της Αμερικανικής Υπηρεσίας Διεθνούς Ανάπτυξης. Κυρίως διακόμασταν από την Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Υπάρχει όμως η διπλωματική πολιτική και υπάρχει και η αναπτυξιακή πολιτική που είναι διαφορετικό το ένα από το άλλο. Εσείς λοιπόν που έχετε τώρα την ε, συνθήκη της Λισαβόνας, έχετε την ε, τρόπο Άστον που είναι αρμόδια αυτά τα θέματα, δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύπλοκο να καταλάβετε ότι υπάρχει μια ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική ε, με την οποία θα πρέπει να είναι συνεπής και η αναπτυξιακή σας πολιτική. Αλλά η αναπτυξιακή πολιτική πρέπει να αποφασίζεται από αυτούς οι οποίοι κατανοούν πώς μπορεί κανείς να πετύχει την ανάπτυξη. Οι μηχανισμοί λοιπόν συντονισμού πιστεύω ότι θα δείτε ότι είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τον κύριο Άτχουντ για μια πολύ σημαντική παρουσίαση και γιατί επίσης έκανε τη διάκριση ανάμεσα στην ανάπτυξη και την εξωτερική πολιτική. Είναι μια διάκριση την οποία αυτή εδώ η Επιτροπή υπογραμμίζει συνεχώς και διευκρινίζει συνεχώς το Κοινοβούλιο. Αλλά βέβαια υπάρχει ένας λευκός ελέφας σε ένα άλλο μέρος του κτηρίου αυτού, τον οποίο δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Γκέι Μίτσελ. Ευχαριστώ τον κύριο Άτχουρ για την παρουσίασή του. Πράγματι δεν είναι πολύ εντυπωσιακή όλοι αυτή οι 13 στόχοι τι συνέβη, γιατί δεν πετυχαίνουμε τους στόχους αυτούς, ποιο είναι το πρόβλημα, ε, ποια είναι τα σημεία τα οποία θα πρέπει να προκαλέσουν την παρέμβασή μας για να υπάρξει βελτίωση. Σε μια τέτοια συνάντηση ίσως ο Φρίτμαν ε, δεν είναι ο κατάλληλος και είχε αναφερθεί στο Freedom to Choose, ε, στο Belmont Syndrome, στο σύνδεδο του Belmont. λέγεται εκεί ε, σε αυτό το κολέγιο στο Μπέλμον ε, μια ολόκληρη σειρά οι καθηγητές έκαναν λάθη στην, στα οικονομικά μέτρα τα οποία πρότειναν διότι ακριβώς ο ένας ακολουθούσε αυτά τα οποία έκανε ο άλλος μόνο και μόνο για λόγους αδράνειας δηλαδή. Ίσως λοιπόν αυτό να φταίει και σε μας. Τώρα να μιλήσω για την οικονομία, την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα. Πράγματι τα εμβόλια τα αγοράζουμε στην καλύτερη τιμή σε σχέση με την ποιότητά τους, η αποτελεσματικότητα. Αν ας πούμε από ένα εμβόλιο βγάζουμε 10 δόσεις, θα βγάλουμε 10 δόσεις. Και η αποτελεσματικότητα επίσης με άλλο τρόπο είναι αν έχουμε πετύχει ας πούμε ε, τους στόχους για την, 90 για την παροτίτιδα. Έχουμε πετύχει τους στόχους μόνο κατά 75 με 80 περίπου τις 100. Οι διαδικασίες όπως είπατε είναι πολύ περίπλοκες και τι μπορούμε να κάνουμε για να τις ελαφρύνουμε τις διαδικασίες αυτές, τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε μεγαλύτερη όμως δυνατότητα αναγνώρισης ευθύνης. Θα πρέπει τους στόχους αυτούς να τους ξεπεράσουμε. Εσείς πηγαίνετε καλύτερα από μας και πόσο και σε ποιους τομείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο Ρικάρντο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τον κύριο Άτογκοτ που είναι μαζί μας σήμερα εδώ. Θα ήθελα δύο ερωτήσεις να υποβάλω. Η μία σχετίζεται άμεσα με την τριαδική, τριγωνική συνεργασία και την συνεργασία νότου-νότου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει να είναι ένας πρωταγωνιστής και όλο και μεγαλύτερο ρόλο θα δραματίσει πιστεύω και στο μέλλον στην ε, συνεργασία αυτή, νότου-νότου και στην τριγωνική συνεργασία. Ξέρετε ότι υπάρχουν αναπτυγμένε χώρε που χρησιμοποιούν αυτή τη βοήθεια. Η Ιαπωνία, που είναι ο ηγέτη ε, στην ε, τριγωνική συνεργασία, συνεργασία νότου-νότου. Ένα αυτό. Ποια είναι η άποψή σα. Δεύτερον, η χρηματοδοτική βοήθεια είναι ένα θέμα που έχει έχουμε εμεί αρμοδιότητα γι' αυτό στην Επιτροπή μα, Η ατζέντα, το θεματολόγιο, λόγω της οικονομικής ε, κρίσης ε, έχει ως αποτέλεσμα θέματα εγκάρσια πολύ σημαντικά να τα βάζουμε σε δεύτερο πλάνο. Κλιματική αλλαγή είναι ένα πολύ σαφές παράδειγμα. Παρότι είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα, δυστυχώς έχουμε αυτή την οικονομική κατάσταση που ε, έχει αυτά τα αποτελέσματα. Κάθε μέρα όλοι μας νομίζω παίρνουμε αναφορές από την ΕΚΟ, την Υπηρεσία Ανθρωπιστικής Βοήθειας, σε σχέση με φυσικές καταστροφές κυρίως που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Έχω λοιπόν ένα σχετικό ερώτημα. Στο περιθώριο της δεσμευσής μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση, τι παγκόσμια δέσμευση βλέπετε να υπάρχει σε σχέση με τη κλιματική αλλαγή και γενικότερα με την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Ευχαριστώ Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να χαιρετήσω την παρουσία του κυρίου Άτχουντ σχετικά με τον ΩΣΑ και την προσπάθεια την αναπτυξιακή που κάνει έχουμε να κάνουμε με έναν εταίρο πάρα πολύ σημαντικό. Είστε εσείς οι οποίοι μας διαβεβαιώνετε ότι τα χρήματα τα οποία εξοδεύουμε στην ανάπτυξη ε, πράγματι ε, δεν πηγαίνουν χαμένα. Ταυτόχρονα ο Σά έχει δημιουργήσει ένα σύστημα αξιολόγησης σε σχέση με την αποτελεσματικότητα, τη διάρκεια ε, γενικά μια ολόκληρη σειρά από στόχους οι οποίοι μας διαβεβαιώνουν για τη σωστή πολιτική που ακολουθούμε. Αναφερθήκατε σε ένα θέμα σημαντικό, την συνεκτική, τη συνεκτικότητα των πολιτικών μας χώρες όπως η Νορβηγία και η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία σαν παράδειγμα αμφισβητεί τη συνοχή της πολιτικής μας στιγματίζοντας κυρίως την ΚΑΠ. Μπορείτε να είστε επακριβέστερο σε ποιο βαθμό η ΚΑΠ μπορεί να βλάψει τις υποανάπτυξη χώρες, γιατί έχουν πλέον οι επιδοτήσεις της εξαγωγής σχεδόν εξαφανιστεί. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό το οποίο ονομάζω η ικανότητα να δίνουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα, να κερδίζουμε συγκριτικά πλεονεκτήματα μέσω της ε, αναπτυξιακής μας πολιτικής. Από τη μία θα πρέπει να υπάρξει αξιολόγηση της πολιτικής συνεργασίας της Ένωσης και από την άλλη μια αξιολόγηση θα έλεγα ε, της δράσης των άλλων, των ΙΠΑ, της Ινδίας κτλ. Υπάρχει μια τέτοια σύγκριση ή μήπως θα πρέπει να εφεύρουμε την μεθοδολογία η οποία απαιτείται για να καταλήξουμε ε, στο να υπάρξουν και κάποια συγκρινικά πλεονεκτήματα από κάποιες πολιτικές. Αν υπάρχει αυτή η δυνατότητα λοιπόν, μπορείτε να μας πείτε πώς μπορούμε να ξεκινήσουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Ένα τελευταίο στοιχείο. Κάνατε μία παρατήρηση με την οποία συμφωνούμε από τότε που ξεκίνησε η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τη θέση σε ισχύ της νέας συνθήκης. Είπατε ότι με νέες μορφές ε, συνδυαστικές η αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να καθοριστεί πλήρως από ε, ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά την ουσία της πολιτικής αυτής. Έχετε κάνει κάποιες ε, παρατηρήσεις οι οποίες σας επιτρέπουν να αμφισβητήσετε την ικανότητα της Ευρώπης να λειτουργήσει προς την κατεύθυνση αυτή. Um, Κύριο Μπέρμαν, ευχαριστώ κύριε Άτχοντ που είστε εδώ. Το Κοινοβούλιο έχει κάποιες δυσκολίες στον τρόπο ελέγχου της αποτελεσματικότητας των πολιτικών μας. Δεν είμαστε στις, στις υποανάπτυξη χώρες, δεν είμαστε παρόντες ε, δεν έχουμε τις δυνατότητες που είχατε εσείς στα πλαίσια του peer review το οποίο είχατε κάνει, της αξιολόγησης μέσω ομολόγων. Και φαίνεται ότι το peer review της DAC σημειώνει ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος. Λέγει ότι υπάρχει καλύτερο συντονισμός ανάμεσα στα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν παράδειγμα. Και αυτό είναι καλοδεχούμενο. Αλλά δεν αναφέρει πάρα πολλά και αυτά τα βγάζω από μια βιαστική ανάγνωση. Η έκθεση αυτή δεν αναφέρει και πάρα πολλά, λοιπόν, για το περιεχόμενο των πολιτικών, για τις επιλογές οι οποίες έχουν γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν παράδειγμα, και θα μπορούσατε να είσαστε λίγο πιο συγκεκριμένος εδώ για την ατζέντα για την αλλαγή, την είδατε την ατζέντα αυτή, και ποια είναι άραγε η αξιολόγηση του ΝΤΑΚΟΣΑ για την ατζέντα αυτή και για τις νέες προτεραιότητες οι οποίες έχουν δοθεί στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικότερα. Και ποια είναι η αξιολόγηση που κάνετε εσείς για τις επιλογές αυτές σε σχέση με το τι θεωρεί ο Σαντακ τα ισχυρά σημεία ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δωρήτριας, ως της μεγαλύτερας μάλιστα δωρήτριας ε, ε, περιοχής και πού ακριβώς η ατζέντα για την αλλαγή εντάσσεται και παράγει προστιθέμενη αξία για την Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύοντας τους σωστούς στόχους την οικονομική ανάπτυξη του αναπτυσσόμενου κόσμου, την αντιμετώπιση και μετρίαση των κλιματολογικών συνεπειών, τον εκδημοκρατισμό, τη στήριξη ε, της δημοκρατίας σε όλες τις υπήρους για να αφαιρθώ σε κάποια επιμέρους θα έλεγα σημαντικά πλαίσια. Λοιπόν, μπορείτε να σχολιάσετε λίγο περισσότερο. Και σε σχέση με την εξωτερική πολιτική να πω ότι οι εξωτερικές πολιτικές και οι αναπτυξιακές πολιτικές τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε εκεί ε, στον τομέα αυτό είναι ακριβώς το τι γίνεται σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής. Ε, εδώ κάποια στρατηγικά συμφέροντα μας έχουν παρεμποδίσει στο να είμαστε αποτελεσματικοί στον τομέα της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σμιτ, διευθυντής από την Γενική Διεύθυνση ΔΕΦΚΟ να πάρει το λόγο και μετά θα ζητήσω από τον κύριο Άπκουτ να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Χαίρομαι που σας βλέπω ξανά. Ευχαριστώ που έχετε τονίσει ότι η ομάδα μας έκανε μία πολύ δίκαιη αξιολόγηση και είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε όλες τις συστάσεις και να τις εφαρμόσουμε. Δεν θα αναφερθώ εις ε, τον κατάλογο των θετικών σημείων που έχω στην αξιολόγηση διότι νομίζω ότι η παρουσίασή σας ήταν πολύ σωστή ε, σε σχέση με την προηγούμενη αξιολόγηση που είχαμε κάνει το 2007 και θέλω να απαντήσω στα σχόλια των Ευρωβουλευτών. Ο κύριος Κόρτες ε, ε, έκανε μία ερώτηση και βλέπουμε ότι πρέπει να συνεργαζόμαστε καλύτερα με, στην, ε, με τους συναδέλφους στη Γενική Διεύθυνση ΕΚΟ διότι όπως ξέρετε εξετάζουμε τις κλιματολογικές αλλαγές, την διατροφική ασφάλεια στο στο κέρας της Αφρικής και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα πρώτο βήμα για να υλοποιήσουμε όλα αυτά που μας ζητήσατε στην αξιολόγηση. Δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να προωθήσουμε τις κλιματολογικές αλλαγές και τα κράτη-μέλη να συμβάλλουν ε, στην ε, ε, υιοθέτηση του προγράμματος και να το χρηματοδοτήσουν. Όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Γκέρενς για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ευρωπαϊκής Αναπτυξιακής Βοηθείας, βλέπετε ότι ε, έχουμε σημειώσει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι πρέπει να είναι υπόλαγα τα κράτη για τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στο Μοντερέι και αυτό λειτουργεί σωστά και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε όσον αφορά την σεξουαλική εμπειρία. Ε, πρέπει να λύσουμε στην ΤΕΦΚΟ διάφορα θέματα συγκεκριμένα και δύσκολα, διότι εμείς ε, θα ασχοληθούμε ε, κατά τομείς. ασχολούμε σε έναν βασικό τομέα της ΔΕΦΚΟ και Έχουμε ε, έξι ή εφτά γιατρούς που ασχολούνται ε, στον τομέα μας. Είναι δύσκολο να προχωρήσουμε με 5, 6, 7 άτομα και θα πρέπει να προσελκύσουμε εξωτερικούς εμπειρογνώμονες ε, που να έχουν τις κατάλληλες ε, γνώσεις και αυτό είναι κάτι που έχει αποδεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν μπορούμε όμως να εστιαστούμε σε λιγότερους τομείς θα είναι πιο εύκολο να προωθήσουμε το θέμα αυτό. Μετά, όσον αφορά τον κύριο Μπέρμαν, δεν αναφερόμαστε στις αλλαγές που έχουν γίνει στην ε, ε, ε, ε, στην ε, ε, ατζέντα για την αλλαγή, Agenda for Change και πρέπει να σας πω ότι η Agenda for Change ουσιαστικά παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και ως εκ τούτου η αναθεώρηση την οποία κάναμε και ε, η ενημέρωση δεν αναφέρεται τόσο με αυτά τα θέματα απλώς ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι στο επίκεντρο αυτής της αλλαγής και αυτό είναι που ο, μας απασχόλησε περισσότερο. Μετά, ο συνδυασμός μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής ε, και της συνεργασίας. Βέβαια, πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι, δεν πρέπει να το λέω έτσι ίσως, αλλά αυτό που προσπαθούμε από δικιά μας πλευρά είναι να, χρησιμοποιήσουμε τους συναδέλφους όχι σαν εχθρούς αλλά σαν ε, φίλους οι οποίοι μπορούν να μας βοηθήσουν να προωθήσουμε τους αναπτυξιακούς στόχους μας. Σαν παράδειγμα θα σας πω ότι δεν μπορούμε να έχουμε επιτυχής διαπραγματεύσεις στις ε, συζητήσεις αυτές αν ε, δεν έχουμε σωστή ενημέρωση σχετικά με την πράσινη ανάπτυξη. Δηλαδή ε, μόνο έτσι θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τις οικονομικές επιπτώσεις εξού και υπάρχει μία υπηρεσία ε, και συνεργαζόμαστε με την υπηρεσία αυτή σε αυτό το πνεύμα. Ε, θα σταματήσω εδώ και πάλι θέλω να πω ότι για μας πρόκειται για μία μεγάλη βελτίωση. Κάναμε αυτά που υποσχεθήκαμε τα τελευταία χρόνια και για τις συστάσεις αναγνωρίζουμε ότι ακόμη μένουν πολλά να γίνουν για την απλοποίηση των διαδικασιών, για την ε, κοινοποίηση των αποτελεσμάτων. Αυτά τα θέματα είναι προσυζήτηση για την επόμενη δημοσιονομική περίοδο και σας ευχαριστώ. Λοιπόν, νομίζω ότι τώρα έχετε πολλά να κάνετε, λέει ο πρόεδρος τον ε, κύριο Άτγουτ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αλλά με εντυπωσίασαν πολύ τα ερωτήματα και πολλές φορές όταν μιλάω στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών περιμένω τέτοιες ερωτήσεις, δεν το περίμενα όμως εδώ και συμφωνώ με το τελευταίο σχόλιο ότι υπήρξε σημαντική πρόοδος όχι μόνο από την τελευταία αναθεώρηση αλλά και στις διμερείς ε, συζητήσεις που παρακολουθώ από τη δεκαετία του 1990 με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπουμε ότι οι πρώην διπλωματικοί ε, ανελάμβαναν την απόστα και δεν θέλω να είμαι αρνητικός εδώ αλλά πιστεύω ότι και εγώ ε, ήμουν, ε, ερχόμουν από το ίδιο, από την ίδια προέλευση, δηλαδή ήμουν ένας διπλωμάτης στο παρελθόν. Ε, αντιλαμβάνεστε, δεν υπάρχει κανείς τέλειος και γι' αυτό δεν πρέπει να κατακρίνω. Αλλά το πιο βασικό ήταν η αξιολόγηση των ε, ομολόγων μας και βλέπαμε ότι οι διπλωματικοί στόχοι πολλές φορές ήταν ε, ε, βραχυπρόθεσμοι και αυτό δεν βοηθάει στη διαχείριση των πόρων. Ε, ε, δηλαδή έπρεπε να ξέρουμε τι μέλη γενέστε ε, σε, για ένα πρόγραμμα με μια προοπτική 20 ετίας και πολλές φορές πρέπει να δούμε και να αξιολογήσουμε αν πρέπει να επιζητήσουμε με τους πόρους βραχυπρόθεσμα διπλωματικά ωφέλη ή μακροπρόθεσμα ωφέλη από την εφαρμογή μιας επικοδομητικής πολιτικής και όλα αυτά περιλαμβάνονται στην Agenda for Change όπου υπάρχει και μία διαφοροποίηση για ένα θέμα που προανέφερα ότι δηλαδή ε, πρέπει να υπάρχει ισότητα και αυτή πρέπει να αντικατοπτρίζεται και στις δηλώσεις ε, για να μπορέσει να δοθεί το σωστό μήνυμα παντού. Πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχει μία συζήτηση για το εάν στο Μπουσάν θα πρέπει να βασιστούμε σε μία μεθοδολογία που να προωθεί τα δικαιώματα διότι κατά τα άλλα προωθούμε την κοινωνία των πολιτών, τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων στην αναπτυξιακή διαδικασία και ε, πρέπει να υπάρχει ε, μία ανάπτυξη η οποία να μας βοηθήσει και γι' αυτό πιστεύω ότι αυτό είναι ε, κάτι πολύ σημαντικό και ε, όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ε, γιατί επιτύχαμε μόνο ορισμένους από τους ε, στόχους μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ένα ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον και βλέπουμε ότι υπάρχει το το πρόγραμμα Erasmus το οποίο δίνει δωρεάν υποτροφίες δεν θα υλοποιηθούν ίσως μέχρι το 2015 είναι όμως ρεαλιστικό αυτή τη στιγμή να πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις υποτροφίες προς τους φοιτητές του τρίτου κόσμου για να ε, ε, ε, για να σπουδάσουν στην Αμερική εάν παράγουν οι χώρες αυτές πάρα πολλά τρόφιμα πιστεύετε ότι έτσι θα ανοίξουν τις αγορές τους πιστεύω ναι διότι αυτές θα καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο χώρο των συναλλαγών και υπάρχουν και πολιτικές πτυχές που καθιστούν δυσχερές να ε, διαφοροποιήσουμε την ε, βοήθειά μας. Υπάρχουν πολλοί ε, οι οποίοι δεν είναι ικανοποιημένοι με αυτό διότι θέσαμε σαν ορόσημο το 2015 και στο παρελθόν είχαμε αναρωτηθεί αν μπορούμε να δώσουμε ε, πληροφορίες για την επόμενη πενταετία στους ομολόγους μας ε, έστω και υπό προϋποθέσεις. Ε, δεν είμαι βέβαιος ότι είναι σωστό αυτό, αλλά ξέρω ότι πολλές χώρες ακολουθούν αυτή την οδό και ζητούν από την εκτελεστική αρχή να προτείνουν στο Κοινοβούλιο ότι ξέρουν ποια κατεύθυνση θα ακολουθηθεί και πολλές φορές οι πληροφορίες αυτές ε, δεν διατίθενται ακόμη στις υποανάπτυξη χώρες. Αλλά τώρα έχουμε προοδεύσει διότι 90% των προβλέψεων αυτών μεταδίδονται στο DAC και το 75% των μελών του DAC λέγουν ότι δεν μας ενοχλεί να το δημοσιοποιήσετε. Εκεί πρέπει να προχωρήσουμε για να καλύψουμε τους στόχους του 2013 αλλά βλέπετε ότι ακόμη δεν έχουμε δεχθεί την πολιτική πραγματικότητα που λέγει ότι χρειαζόμαστε αυτά αποτελέσματα και αυτό είναι το πιο σημαντικό διότι αν δεν το δεχθούμε θα έχουμε δυσκολίες να καλύψουμε τις υποχρεώσεις μας και το θέμα δεν είναι οι αναπτυξιακές οι αναπτυξιακές ε, ε, ε, οργανώσεις που εξαρτώνται από τη συνεργασία με τους ομολόγους τους αλλά το ευρύτερο κοινό και ίσως γι' αυτό μέχρι τη στιγμή δεν πετύχαμε τους στόχους μας το Μπουσάν είναι πολύ σημαντικό και ε, όσον αφορά την ερώτηση για τις κλιματολογικές αλλαγές και τις φυσικές ε, καταστροφές ε, και τους ε, αντιχτύπους τους που έθισε ένας από τους κυρίους πρέπει να σας πω ότι καταρτήσαμε την πρώτη έκθεση όπου λέμε πόσα ξοδεύουμε για τις προσαρμογές που χρειάζονται από τις κλιματολογικές αλλαγές. Οι 22 εκατομμύρια πέρυσι αναφέρθηκαν σε αυτή την προσαρμογή και μόνο 8 εκατομμύρια από τα 22 ήταν ε, ουσιαστική προσαρμογή και θα χρειαστεί να βελτιώσουμε αυτή την επίδοση γιατί θα πρέπει να υπάρχουν προσθετικές συνεργίες και μπορεί να μην είναι το ODA, μπορεί να είναι άλλες ροές που θα καταλήξουν στην κλιματική χρηματοδότηση και είναι θέματα που πρέπει να εξετάσουμε. Ετέθη ένα ερώτημα για την συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ενάσεως με ένα άλλο μέρος του ΝΤΑΚ ε, με την Ιαπωνία, αλλά προτιμώ να μην το σχολιάσω τώρα. Ε, νομίζω ότι κινήσατε το ενδιαφέρον με τα 8 δισεκατομμύρια ή εκατομμύρια. Πού τα βρήκατε. Ξέρετε πού τα βρήκατε. Αυτή είναι πόρη τους οποίους μας ανέφεραν τα μέλη του ΝΤΑΚ. Δηλαδή προέβησαν σε μία ανάλυση για να δουν αν είχαν δαπανηθεί τα προγράμματα αυτά για την προσαρμογή στις κλιματολογικές αλλαγές. Εν μέρει ήταν γεωργικά προγράμματα και μας έδωσαν πολύ συγκεκριμένα λεπτομερή στοιχεία, αλλά δεν μπορώ να σας πω εγώ ακριβώς πώς διετέθησαν και απλώς να σας πω ότι ε, χρησιμοποιήθηκαν εκεί που ήταν πραγματικά αναγκαία. Αναγκαία, okay, ένα σύντομο ερώτημα. Δεν ξέρω αν ήσασταν ε, πιο πριν κυρία αλλά πριν συζητήσαμε εδώ την ανάγκη εμείς ε, να έχουμε από στο πλευρό μας και την κοινή γνώμη με όλα αυτά τα προγράμματα λιτότητας, θέλουμε να υπάρχει αποτελεσματικότητα κτλ. Η πραγματικότητα, η λιτότητα δηλαδή αυτή που αντιμετωπίζουμε. Κάνει πιο ευαίσθητους αυτούς που ηγούνται αυτών προγραμμάτων ε, σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα των πόρων που διατίθενται. Έχετε αυτή την εντύπωση. Απάντηση. Μπορώ να το συγκρίνω αυτό μόνο με τη δεκαετία του 90 όταν προσπαθούσαμε να βάλουμε πλαίσια για αποτελέσματα. Υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γινόντουσαν μετρήσεις, υπολογισμοί. Υπήρχε υποχρέωση να φανεί στους φορολογουμένους ότι υπήρχε αποδοτική χρήση των κονδυλίων. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τώρα είναι να εξασφαλίσουμε οι χώρες εταίροι να μετρήσουν και αυτές διότι υπάρχει ένα πρόβλημα ή καλύτερα μία πρόκληση ε, σε ό,τι αφορά την απόδοση ε, είτε των ευθυνών είτε των ευσύμων ε, για τα αποτελέσματα. Τα επίπεδα της ε, αναπτυξιακής βοήθειας είναι καταλητικά. 130 δις είναι ε, το ποσό αυτό σε δολάρια. Αλλά με τις κυβερνήσεις εργαζόμαστε και θα πρέπει να κινητοποιήσουν αυτές και χωρίς πόρους και να επενδύσουν στην ανάπτυξή τους. Όταν λοιπόν οικειοποιούνται τα προγράμματα, τότε έχουμε αποτελέσματα. Θα πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα συστήματα που θα μπορούμε μαζί οι χώρε αυτέ και εμεί να μετράμε τα αποτελέσματα. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε για τη λιτότητα. Επειδή η G20 επικεντρώνεται στην παγκόσμια οικονομική κρίση, κάποιοι ηγέτε, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επικεντρώνονται ε, πιο πολύ από ποτέ στην ανάπτυξη που γίνεται ένα κεντρικό λίθος τη παγκόσμια πολιτική πολύ περισσότερο από ό,τι παλιότερα. Και Κάποιοι βλέπουν σαν αναπτυσσόμενο κόσμο κάποιε δυνατότητε ανάπτυξη, αλλά υπάρχουν, όπω ξέρετε, στην Δύση ανάπτυξη, ε, δημογραφικά προβλήματα. Έτσι λένε κάποιοι ότι θα πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη. Και πράγματι αυτό ίσως για ανθρώπους που βιώνουν τη λιτότητα να μην είναι εύκολο αλλά νομίζω ότι είναι όλο και πιο πιστικό ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην οποία τη βοήθεια και σε άλλες ροές, ώστε να ενισχύσουμε ε, τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην ανάπτυξη. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος, κύριε Πρέσβη, σας ευχαριστώ. Ο Σάρλ έχει το λόγο. Ο κύριος Σάρλ απάντησε στο ερώτημά μου για το κατά πόσον μπορούμε να τονίσουμε και να προβάλλουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της αναπτυξικής πολιτικής της Ένωσης σε σχέση με άλλα μέλη της ε, ΤΑΚ και είπατε ότι δεν θα απαντήσετε σε αυτό το ερώτημα. Μήπως όμως μπορείτε να απαντήσετε στα άλλα ερωτήματα που σας έθεσα, δηλαδή η σύγκριση μεταξύ της δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνα, για παράδειγμα. Πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι είναι προφανές, αν διαβάσει κανείς και την αξιολόγηση των απομοτήμου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συμβάλλει τα μάλα, ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στην ανάπτυξη σήμερα ανά τον κόσμο. Η Κινέζη, το κινέζικο πρόγραμμα είναι λίγο σκοτεινό θα έλεγα. Έχουμε κάνει πολλές επισκέψεις εκεί. Ίσως να δίνουν 10 δις δολάρια, αμερικανικά δολάρια ε, βοήθειας που έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει με τα εμπορικά του συμφέροντα. Χάρη όμως ε, στον ε, Πρωθυπουργό άρχισαν να ε, βλέπουν και αυτοί τις επενδύσεις. Κάνουν καλές επενδύσεις και έτσι εξολογούν καλύτερα και τα προγράμματα και μπορούμε και εμείς να εξολογήσουμε καλύτερα. Να δούμε, είναι βιώσιμα τα προγράμματα, επιτυγχάνονται αναπτυξιακοί στόχοι. Φαίνεται ότι έχουν αυτό το στόχο και την προθυμία οι Κινέζοι. Υπάρχει και για πρώτη φορά η Λευκή Βίβλος που και λένε στον κόσμο ότι έχουν ένα πρόγραμμα ξένων, ε, ξένης βοήθειας. Και έτσι μπορούν να δείξουν ε, στον κόσμο, στον πληθυσμό της χώρας τους, ότι δαπανούν τα χρήματα με καλό τρόπο. Η ΝΤΑΚ έχει διάλογο, έχουμε την ε, ομάδα μελέτης ΝΤΑΚ Κίνα στα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Ε, ανταλλάξαμε λοιπόν απόψεις μεταξύ τους και πιστεύουμε ότι υπάρχει ελπίδα για μεγαλύτερη τριγωνική συνεργασία. Είναι μια διαδικασία εκμάθησης και επιμερισμού βέβαια των βαρών. Όλοι μπορούμε να μάθουμε ένας από τον άλλο και νομίζω ότι κάνουν ό,τι μπορούν, ε, ίσως περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα για τη μείωση της φτώχειας. Και έχουν εισαγράγει μεθόδους που ούτε εμείς έχουμε στη διάθεσή μας. Ίσως γιατί χρειάζεται να έρθουν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να εξηγήσουν γιατί έκαναν ό,τι έκαναν και τι έκαναν απλά στο Κομμουνιστικό Κόμμα, στην αρχαία του Κομμουνιστικού Κόμματο πρέπει να τα αιτιολογούν, που αυτή τη στιγμή ομφαλοσκοπεί από ό,τι φαίνεται. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ γιατί απαντήσατε με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Γρήγορο ερώτημα. Υπάρχει διάκριση μεταξύ αυτών που εμεί κάνουμε και αυτών που κάνουν άλλοι. Ότι εμείς δηλαδή ίσως καθαρίσαμε κάτι που ε, μάλλον αποσυνδέσαμε. Ε, ναι, η αποσύνδεση και η σύνδεση είναι ένα θέμα. αν έχετε ανοιχτά συστήματα διαγωνισμών, υπάρχει χαμηλότερο κόστος. Αν μπορεί ο καθένας να υποβάλει υποψηφιότητα, αυτό έχουμε αποδείξει. Δεν ξέρουμε πολλά για το κινέζικο πρόγραμμα, αλλά αυτό είναι περιορισμένο. Πράγματι, με τα δικά του συμφέροντα. είναι μέλος της DAC. Πρόοδος υπάρχει. Thank Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ καλή συνεδρία. Σας ευχαριστούμε. Ah, Ολοκληρώνουμε την πρωινή μας συνεδρίαση και θα επανέλθουμε στις 3 ακριβώς, στην ίδια αίθουσα.